Uh, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το τέταρτο τμήμα της συνεδριάσεώς μας, με χαρά. Ερχόμαστε για να συζητήσουμε ένα πολύ συναρπαστικό θέμα, στρατηγική για το διάστημα της Ευρώπης. Και καλώς ορίζω τους ομιλητές μας. συντονιστές ουσιαστικά κήρυξαμε την έναρξη αυτή τη στρατηγική στη χθεσινή μα συνεδρίαση. Στην επίσημη εκδήλωση με τον Αντιπρόεδρο Σεύτσοβιτ και την Επίτροπο Βενιτικότσικα και τώρα και αυτό αποτελεί τη συνέχεια τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέθηκε πριν από δύο εβδομάδε. Νέα ιδέα λοιπόν. 26 Οκτωβρίου δημοσίευσε τη στρατηγική για το διάστημα τη Ευρώπη, της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η στρατηγική έχει σε στόχο να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τη θέση που τη αρμόζει στην έρευνα στο διάστημα, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στην αγορά του διαστήματος να αντλήσει τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη των δραστηριοτήτων των σχετικών με το διάστημα σε ένα βέβαια περιβάλλον ταχύτατα εξελισσόμενο και μεταλλασσόμενο με ταχύτατα εξελίξει στην ε, αγορά και το χώρο του διαστήματος εν γέννη. Και δεν είμαι βεβαίω εάν έχει όντως ηγετική θέση η Ευρώπη προκειμένου να ε, επιβεβαιώσουμε τη θέση μας πρέπει να είμαστε και πρωτοπόροι. Είμαστε λοιπόν, είμαστε, έχουμε ηγετική θέση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση προς τους ομιλητές μας. Γιατί λέγεται με τη στρατηγική ότι θέλουμε να προαγάγουμε ε, την ηγετική μας θέση, πως πρέπει πρώτα να την εξασφαλίσουμε. Έχει δύο ψηφίσματα υιοθετήσει από τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς την καταγραφή, το uptake και δεύτερον τις ευκαιρίες και δυνατότητες για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια σε συνδυασμό με το διάστημα. Δύο τμήματα έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή μας, για την απόψη μας συνεδρία, με δύο μιλητές στο κάθε τμήμα. Και παρακαλώ τους ομιλητές οι δυνατόν να μην ξεπεράσουν το δεκάλεπτο στην ομιλία τους ο καθένας, γιατί προτιμούμε να έχουμε πάντα τη συζήτηση, βεβαίως αν ε, αποδειχθεί απαραίτητο ή κάποια παρουσίαση με τις διαφάνειες χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ίσως είναι αναγκαίο να δώσουμε περισσότερο χρόνο. Στο πρώτο τμήμα λοιπόν, ο μιλητής μας, ο κύριος Ντεσδορίδες, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το διάστημα. Είστε λοιπόν υπεύθυνο αυτή τη υπηρεσία, άρα αρμόδιο για συγκεκριμένε δράσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα θέλατε να μα πείτε, ξεκινώντα, άλλη μια ερώτηση προ εσά, κύριε Διευθυντά. Πώς διαμορφώνεται η δικτύωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής και των Εθνικών Υπηρεσιών Διαστήματος, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ε, αυτά που προτείνεται. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τη δικτύωση, τη διάρθρωση μεταξύ των υπηρεσιών. Πώς είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ποιες χώρες έχουν εθνικές υπηρεσίες και συναφή θέματα. Πέραν όλων των άλλων που έχετε προβλέψει τη διαφανία σας. Και έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση να σας παρουσιάσω αυτό που κάνουμε. Την πρώτη ερώτηση θα την απαντήσω μέσα από τις διαφάνειές μου, αν η Ευρώπη είναι στην πρώτο καθεδρία. Για τη δεύτερη και τη γενικότερη εικόνα. Είμαστε ρυθμιστική υπηρεσία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε στο Συμβούλιο μας τα 28 κράτη-μέλη συν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιδιαίτερα αφιερώνουμε το έργο μας στο GNSS, το Γαλιλαίο και το Γνώσο. Δεν ασχολούμαστε με το κάθε τι δηλαδή στο χώρο του διαστήματος. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Υπογράφουμε τώρα μια πολύ σημαντική συμφωνία. Θα δείτε από τις διαφάνειές μου, αλλά σας το περιγράφω με λίγα λόγια, ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος έχει αναλάβει την ανάπτυξη του συστήματος, ενώ εμείς προσφέρουμε την υπηρεσία. Ένα εγχείρημα μοναδικό, δηλαδή, γιατί είμαστε η μόνη υπηρεσία η οποία εστιάζεται στην προσφορά υπηρεσίας σχετικής με την προαγωγή της αγοράς. και νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες χάρη στην παρουσίασή μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με την πρώτη διαφάνεια που συνιστά μια προσπάθεια να σας εξηγήσω τι κάνει η υπηρεσία μας μέσα από τους τέσσερις βασικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το διάστημα που είναι το θέμα της σημερινής σας συνεδρίασης. Από, τέσσερις, από τις τέσσερις βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας θα δείτε νομίζω αυτό που πράττουμε, αυτό που κάνουμε και είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να εξηγήσουμε σε τι εστιάζουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη αγοράς και ασφάλεια αυτήν οι τέσσερις τομείς. Και ξεκινώ με τον πρώτο άξονα τη στρατηγικής για το διάστημα, μεγιστοποίηση των ε, ε, κερδών, των πλεονεκτημάτων από τη... σε σχέση με το διάστημα για την κοινωνία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Τι κάνει η υπηρεσία μας στο προκείμενο. Δεν έχω τόσο χρόνο, γι' αυτό θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχάς για το έγνος, που είναι πρόδρομος του Γαλιλαίου. Σήμερα Ύστερα από τέσσερα χρόνια δουλειά έχουμε 200 αεροδρόμια που αξιοποιούν το έγνος στην Ευρώπη και χώρες όπως η Γαλλία που ήδη έχουν αναπτύξει σχέδια για την κατάργηση της υποδομής εδάφους που έχουν προς όφελος του έγνος, των υποδομών του έγνος των διαδικασιών του έγνους. Πολύ σημαντικό επιτεύγμα. Δεύτερο σημαντικό επιτεύγμα. Αρχίζουμε και βλέπουμε μια σημαντική ε, ελκυστικότητα του Γαλιλαίου Εφέτος τον Ιούλιο είδαμε ένα πρώτο ευρωπαϊκό τηλέφωνο Made in Europe, πλήρως συμβατό με το σύστημα Γαλιλαίος. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό, διότι δίνει μαρτυρία και για το ενδιαφέρον που δείχνει η αγορά για το σύστημα Γαλιλαίους και το έγνος. Τι κάνει η υπηρεσία μας. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες τάσεις τεχνολογικές, κρίσιμες προκλήσεις και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μία πολύ σημαντική, την αυτόνομη οδήγηση, την οποία είδαμε σιγά σιγά να αναπτύσσεται ε, σε σχέση με το μέλλον του αυτοματοποιημένου απολύτως ε, αυτοκινήτου θα έχουμε βέβαια τη χρήση του GSS, GNSS αλλά όχι μόνο και συνεργαζόμαστε με τους κύριους βιομηχανικούς ε, παράγοντες για την ανάπτυξη του απολύτως αυτονόμου αυτοκινήτου για το μέλλον. Για το δεύτερο πυλώνα και την προαγωγή μιας ε, συνολικά ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής βιομηχανίας για το διάστημα. Έχουμε μια μακρά εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, περί τα 100 έργα του 7ου προγραμμάτος πλαισίου και ε, αρκετά τώρα με το πρόγραμμα έως το 2020. Εφαρμογές και υπηρεσίες πάνω απ' όλα εντάσσονται εδώ και είναι πολλές οι ενδιαφέρουσες ιδέες τις οποίες καλλιεργούμε και προσφέρουμε βοήθεια στους νέους επιχειρηματίες για να μπουν σε αυτήν την πολλά υποσχόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένας άλλος πολύ σημαντικός ρόλος για την υπηρεσία είναι ο ρόλος του καταλήτη, δηλαδή ε, επιτρέπει να κλειδώσουν μεταξύ τους διαφορετικές δεξιότητες ή ρόλοι, ε, οι λειτουργίες, παράδειγμα η πολιτική αεροπορια πορεία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, που δεν υπήρχε τίποτα, ξεκινήσαμε από το μηδέν και μπορέσαμε με πιστοποιημένα ε, διαπιστευμένα όργανα, ε, αεροδρόμια, ε, παρόχους υπηρεσιών, βιομηχανία που τους φέραμε όλους σε επαφή και συνδέθηκαν μεταξύ τους να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και όπως σας είπαμε το έγνος ε, που τώρα χρησιμοποιείται σε πολλά αεροδρόμια του κόσμου έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Για το μέλλον τι σκοπεύουμε να κάνουμε, συνεχίζουμε βεβαίως ε, την ε, δουλειά μας με βάση το Horizon 2020, πολύ χρήσιμο εργαλείο. Έχουμε και άλλα εργαλεία, αυτά που ονομάζουμε θεμελιώδη στοιχεία και αποτελούν εστίαση, σημείο εστίασης της έρευνας και ανάπτυξής μας για την ε, προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και επίσης συνεργασία με τις δημόσιες αρχές όταν αυτές το ζητούν όταν ζητούν δηλαδή υποστήριξη από πλευρά μα για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων, των ε, τυπικών απαιτήσεων ε, ή τεχνικών καλύτερα απαιτήσεων για τα ε, νέα του συστήματα. Εμείς καταγράφουμε όταν μας το ζητούν δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία που χρειάζονται τα τεχνικά δελτία. Και αυτό και για τα νέα οδικά συστήματα που χρησιμοποιούν το νέο GNSS. Τέταρτο σημαντικός πυλώνας είναι η ενίσχυση της ε, αυτονομίας της Ευρώπης στην πρόσβαση και στη χρήση του περιβάλλοντος σε ένα ασφαλές χωρίς κινδύνους περιβάλλον. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από το GNSS, το οποίο έχει πια ε, μπει στην καθημερινή μας ε, ζωή και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έχει σημεία ευάλωτα το GNSS και άρα η διάσταση της ασφάλειας παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία Και εδώ θέλω να τονίσω προς εσάς το γεγονός ότι το Genesis αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους κύριους παράγοντες εξασφάλισης της ασφάλειας. Στο χώρο του διαστήματος έχουμε 30, ε, μια υπηρεσία 30 ατόμων στη Γαλλία, στο Παρίσι, εκ των οποίων 20 είναι από τη δική μας ε, η υπηρεσία δουλεύουν ε, επί 24 ώρου βάσεως στην ανάπτυξη του τμήματος που ονομάζουμε PRS User, δηλαδή αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν το κρυπτογραφημένο μήνυμα για χρήση στην αγορά, με μια ειδική τεχνολογία που φυσικά δεν είναι διαθέσιμη στην εμπορική αγορά. Και, εν τέλει πολύ σημαντικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ε, υπηρεσία μας πιστοποιεί τις απαιτήσει ασφαλείας. Ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Η υπηρεσία μας όμως προσφέρει την πραγματογνωμοσύνη, τις τεχνικές γνώσεις για να ε, αξιολογηθούν οι διάφορες διαστάσεις, τεχνικές διαστάσεις της ε, ασφάλειας του συστήματος. Η τέταρτη διάσταση του συστήματος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και ε, η προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας. Εδώ ο ρόλος της υπηρεσίας μας είναι να συμμετέχει σε διάφορα διεθνή έργα και προγράμματα. Ε, ενεργά προσφέρουμε την υποστήριξή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διεθνείς της δράσεις. Ιδιαίτερα θέλω εδώ να σας πω ότι ήδη λαμβάνουμε πολλά θετικά και υποσχόμενα, πολλά υποσχόμενα μηνύματα. Ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο της προηγούμενης εβδομάδας, ένας, ε, μια βιομηχανική ε, δραστηριότητα που ξεκινάει σε συνεργασία στη Νότια Κορέα με την εφαρμογή του έγνος έχει υπογραφεί σχετική σύναψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για, για, τον, για, την αλόγω επιχείρηση, αλλά πολύ σημαντική ιδιαίτερα για μας γιατί σημαίνει ότι αρχίζει η διάδοση του συστήματος και πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστια η ε, ανταγωνιστική πίεση από τον ανταγωνιστή στι ΗΠΑ. Φυσικά το γνωρίζετε αυτό και το καταλαβαίνετε. Και φτάνω τώρα στη τελευταία μου διαφάνεια, που αφορά κατά βάση μία σύνοψη του ρόλου της έγνος. Βλέπετε εδώ τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών, την ασφάλεια, την ανάπτυξη της αγοράς, τη διαχείριση εφαρμογών και την επικοινωνία και προαγωγή. Δεν κάνουμε απλώς μια απογραφή της κατάστασης, δεν συντάσσουμε εκθέσεις. Έχουμε δραστηριότητα και μοναδική τεχνογνωσία. Και νομίζω ότι είμαστε και μοναδικοί υπ' την έννοια ε, στον κόσμο. Μέσα στα λίγα αυτά λεπτά που είχα στη θέση μου πιστεύω ότι σας έδωσα μια γενική και καλή επισκόπηση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας μας. Μια τελευταία παρατήρηση σχέση με, τις, ε, με τους πόρους μας. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι το πολύ δημοφιλές εν γέννη τον τελευταίο καιρό. Θέλω μόνο να γνωρίζετε ότι ό,τι βλέπετε σήμερα έχει επιτευχθεί με 100 άτομα στο προσωπικό μας που διαχειρίζονται ένα έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1,45 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τελευταία τετραετία. Έχουμε λοιπόν ανάγκη για περισσότερους πόρους. Τις δυσκολίες τις ξεπερνούμε χάρη σε ε, εξωτερικούς συμβούλους ε, υψηλής βέβαια ε, υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας, που βέβαια δεν σημαίνουν πάντα και πολύ οικονομικές λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. 4,5 δισεκατομμύρια. Σωστά. Ναι. Δημόσιας χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020. Σημαντικό ποσό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Μπατιστόν, που είναι πρόεδρος της Ιταλικής Υπηρεσίας Διαστήματος και στο Πανεπιστήμιο του Τορέντο, καθηγητής. Ωραία. Έτσι θα δούμε την κατάσταση και από την πλευρά, από την οπτική γωνία των εθνικών υπηρεσιών διαστήματος. Κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι ρυθμιστική. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της εθνικής άποψης και των εθνικών διαστημικών υπηρεσιών μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική διαστήματος και τις δραστηριότητες της διαστημικές. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Ναι, μου ζητήσατε να έρθω και να συζητήσουμε εδώ για τον ρόλο των εθνικών διαστημικών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το διάστημα στην Ευρώπη έχει να κάνει με την δραστηριότητα τριών οργάνων. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, που συμμετέχουν 22 χώρες, Κάποιες από αυτές, δύο ή τρεις, δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύνολο των εθνικών υπηρεσιών διαφορετικού μεγέθους, σε διαφορετικό πλαίσιο και με διαφορετικές ικανότητες επενδυτικές. Η Ιταλική είναι αυτή που γνωρίζω καλύτερα βέβαια, οπότε αυτά που θα σας πω εφαρμόζονται σίγουρα στην Ιταλία, αλλά ίσως και σε κάποιες άλλες που συμμετέχουν με εθνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν ε, αυτά τα τρία σώματα μεταξύ τους δρούν. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και η Ευρωπαϊκή Ένωση η σχέση είναι κάπως ιδιαίτερη γιατί είναι οι ίδιες χώρες που εδρεύουν γύρω από το ίδιο τραπέζι θα μπορούσαμε να πούμε. Μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις αποφάσεις τους, πώς συνδυάζονται τη στιγμή που πρόκειται για τις ίδιες πηγές πόρων. Είναι ένα δύσκολο θέμα, γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος γιατί αντιμετωπίζει κάποια από αυτά τα προβλήματα. Και μετά κυβερνητικά ε, λογοδοτούν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες διαστήματος. Πρόκειται λοιπόν για έναν μηχανισμό με τρία μέρη. Το θέμα είναι πώς μεταξύ τους συνδέονται αυτά τα τρία μέρη και πώς λειτουργούν μεταξύ τους. Μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα των μεγάλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας Γαλιλαίο, Καπέρνικος, Αμαστή. και βλέπουμε ότι ανάλογα με το πρόγραμμα η σχέση μεταξύ των τριών σωμάτων διαφέρει. Για παράδειγμα για το Γαλιλαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσαμε για το GSA, συζητάμε για υπηρεσίες, μιλάμε για τις εφαρμογές δεδομένων, την ανάπτυξή τους, η να χρησιμοποιήσει η διαστημική οικονομία τα δεδομένα από το Γαλιλαίο και να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί και να μελετήσει και το μέλλον και την εξέλιξη του Γαλιλαίου, πώς θα συνεχίσουμε με αυτό. Αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο από την άλλη μεριά είναι ένα τεχνικό όργανο το οποίο εφαρμόζει τη στρατηγική. Διασφαλίζει ότι μπορούν να φτιαχτούν και να εκτοξευθούν σωστά οι δορυφόροι, ότι θα υπάρξει κοινή διαχείρισή του και φροντίζει και για τι σχετικέ υπηρεσίε. Οι εθνικές υπηρεσίες τώρα ασχολούνται με το PRS, που είναι το τμήμα της ασφάλειας του Γαλιλαίου. Συμμετέχουν σε δράσεις πολλές φορές, φροντίζουν οι υπηρεσίες να εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσουν εφαρμογές και διασφαλίζουν ότι οι εθνικές οικονομίες εποφελούνται από τη διαστημική οικονομία. Αν δείτε τον Κοπέρνικο, εδώ η οργάνωση είναι κάπως διαφορετική μεταξύ των τριών σωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι είναι το όργανο εκείνο, το κύριο στοιχείο του Κοπέρνικου που φροντίζει τα δεδομένα που έχουμε από το δορυφόρο αυτό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο και στην οικονομία. Φροντίζει και για ε, εφαρμογές και πώς θα προωθηθεί σε επίπεδο χωρών μελών και στην Ευρώπη γενικότερα το Κοπέρνικους. Και βέβαια η διαστημική οικονομία είναι το πιο βασικό. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος φροντίζει για δορυφόρους, για δράσεις, για έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά τα δεδομένα και έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά τι εφαρμογές. και φροντίζει να υπάρχουν επιπτώσεις θετικές επί της οικονομίας και ωφέλη για την κοινωνία. Αυτό το κάνουν οι εθνικές υπηρεσίες. Αν δείτε τώρα το SST, που είναι η διαστημική εποπτεία και χνηλάτιση, εδώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές υπηρεσίες. Εδώ πρόκειται για δύο μόνο στοιχεία. Άρα, έχει φτιαχτεί ένα κονσόρτιουμ από τις εθνικές διαστημικές υπηρεσίες για να συζητήσουν τις διάφορες δράσεις να υπάρχει αρκετό κεφάλαιο για να στηριχθεί το consortium. Και εδώ αυτό γιατί το λέω, γιατί δεν υπάρχει ένας ενίος κανόνας για την λειτουργία των τριών αυτών σωμάτων. Ανάλογα με την περίπτωση έχουμε δύο ή έχουμε τρία και η σχέση μεταξύ τους μπορεί να είναι διαφορετική. Τώρα, η στρατηγική, η διαστημική στρατηγική είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η Επιτροπή φρόντισε όλα αυτά τα στοιχεία, οι χώρες μέλη, η ΙΖΑ και τα λοιπά μπορούν ε, να συνεισφέρουν όλοι σε μια συζήτηση που κράτησε βέβαια αρκετό καιρό. Και καταλήξαμε σε αυτό το έγγραφο, το οποίο καθορίζει το τι έχουμε και πού θέλουμε να πάμε προς το συμφέρον της Ευρώπης συνολικά. Νομίζω ότι το γύριμα έγινε καλά. Υπάρχουν οι βασικοί πυλώνες υπέρ της κοινωνίας και της οικονομίας, υπάρχει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υπάρχει η ενίσχυση των προγραμμάτων για, για το διάστημα, υπάρχει ενίσχυση επίσης της Ευρώπης και του ρόλου της ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή. Έχουμε τώρα τα προγράμματα Γαλλία Κοπέρνικος και το SST, αλλά σκεφτόμαστε και τις μελλοντικές εξελίξεις στο GovSatcom, τους εκτοξευτές και το IOV και IOD. Γι' αυτά τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση. Πάντα ακολουθώντα αυτή την λογική που λέει ότι πρέπει να υποφεληθεί η κοινωνία από το διάστημα και χρησιμοποιείται φυσικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος πάντα για τα τεχνικά ζητήματα και οι εθνικές υπηρεσίες διαστήματος φροντίζουν σε επίπεδο χωρών μελών να διαπιστωθούν αυτά το φέλη. Θα πάρω δύο παραδείγματα. Η Ιταλική, για παράδειγμα, υπηρεσία διαστήματος, πώς συνεισφέρει σε αυτό το μοντέλο. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι το διάστημα αλλάζει και αλλάζει πολύ γρήγορα. Αυτή η εικόνα συγκεκριμένα δείχνει ο διαστημικός μας ε, σταθμός, πώς έχει φτιαχτεί, για να εκτοξεύει δορυφόρους, για νέες εφαρμογές, οι οποίες όπως ξέρουμε έχουν ε, αλλάξει τον κόσμο και την παρατήρηση του κόσμου. Το 1971 η Αμερικανική εταιρεία πριν από λίγα χρόνια εκτόξευσε νάνο δορυφόρους με 150 ε, εκατομμύρια κεφάλαιο. Και εδώ έχουμε τη χρήση ε, μιας ενός πυράβλου. Οπότε αυτά είναι δύο παραδείγματα μόνο για το πώς εξελίσσεται το διάστημα τον τελευταίο καιρό και πόσο γρήγορα πρέπει εμείς να αντιδράμε για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις εξελίξεις. Συνεπώς, οι διάφορες υπηρεσίες και η βιομηχανία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αλλαγές και να προσαρμόζουν ανάλογα την πολιτική τους. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια συνεχή ε, διάδραση και σχέση μεταξύ των τριών σωμάτων που σας εξήγησα πριν για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Η διαστημική οικονομία είναι από τα κύρια στοιχεία στη συζήτηση. Είναι ένα νέο είδος οικονομίας που χρησιμοποιεί το διάστημα για ένα πολύ καλό σκοπό. Το διάστημα προσφέρει πολλά στοιχεία και η μελλοντική οικονομία έχει να κάνει με το διαδίκτυο, με την χρήση των δεδομένων και τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες μέσω δεδομένων Έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές στο μέλλον. Άρα πρόκειται για πλούτο, για ωφέλη που μπορούμε να έχουμε και πολύ γρήγορα μάλιστα. Το ερώτημα βέβαια που θέτουμε φτάνουν όσα κάνει η Ευρώπη για να ενισχύσει τη διαστημική μας οικονομία. Τα καταφέρνουμε, είμαστε στο χρόνο μας μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε ε, τα πράγματα ή το σημερινό επίπεδο της χρηματοδότησης. Αν δείτε εδώ τον προπολογισμό, βλέπετε τη συνεισφορά των υπηρεσιών, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Εθνικό Τμήμα δηλαδή, το Ευρωπαϊκό και η Κομισιόν. Έχουμε και τις ΗΠΑ στην Άσα και τη Ρωσία. Εμεί είμαστε κάπου ανάμεσα. Βέβαια εξαρτάται πώ το βλέπει κανείς. Βλέπετε τους κόκκινους κύκλους και αυτοί οι κόκκινοι κύκλοι είναι και η εθνική συνεισφορά και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Κομισιόν. Οπότε εξαρτάται αυτή η κύκλη μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με το αν λαμβάνετε υπόψη σας και τα τρία αυτά στοιχεία ή όχι. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να δούμε. Εμείς είμαστε το σύνολο πολλών και διαφορετικών δράσεων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε καλά συντονισμένοι, να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να μην υπάρχουν κενά για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στην Ιταλία λοιπόν αυτό το κάνουμε. Προσπαθούμε ο μηχανισμός αυτός που έχουμε και σε εθνικό επίπεδο, γιατί και εμείς έχουμε διάφορους φορείς στη χώρα μας που θέλουμε να επωφεληθούν από το διάστημα. Προσπαθούμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο φορέα σε επίπεδο Πρωθυπουργού, ώστε η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία, τα Υπουργεία ή η βιομηχανία να συναντιόνται μεταξύ τους κάθε τόσο, ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάνουμε σωστά την πολιτική μας σε εθνικό επίπεδο. Και τα καταφέραμε, γιατί πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε και η κυβέρνηση για πρώτη φορά αποφάσισε να φέρει φρέσκο χρήμα από ένα ειδικό ταμείο, το τσίπε όπως το λέμε, για στρατηγικές επενδύσεις όσον αφορά τη διαστημική οικονομία. Επιλέξαμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το διάστημα, γιατί ακριβώς πρόκειται για πολλά υποσχόμενη συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα, κυρίως χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Να και ένα παράδειγμα που σας φέρνω για το τι μπορεί να κάνει μια εθνική διαστημική υπηρεσία. Νέες τεχνολογίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Η ίδια Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία μπορεί να φτιάξει υποδομές. Αλλά πρώτα έρχονται οι εθνικές υπηρεσίες με κάποιες ιδέες. Το κόσμος είναι ένα καλό παράδειγμα. Είναι μια υποδομή που έχουμε για διτές, διπλές εφαρμογές. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε στοιχεία και για στρατιωτικές και για μη στρατιωτικές εφαρμογές. Για διαστημική υποπτή και χνηλάτιση ή άλλα. Επειδή λοιπόν το κόσμος και το Sentinel-1 αποφασίστηκε να είναι δορυφόρος, το κόσμος και το Sentinel-1 πρέπει να ξέρετε ότι κάνουν διαφορετικά και συμπληρωτικά πράγματα. Εδώ βλέπετε τη Φλωρεντία. Υπάρχει ένα κομμάτι, σας τα διαβάσατε ε, και σε εφημερίδες, ότι κατέρευσε αυτό το κομμάτι. Έχουμε όμως στοιχεία για σταθερότητα και παληθεύουμε έτσι τι κινείται, τι μετακινείται με αυτή την δορυφορική εικόνα. Και εδώ βλέπετε την ευαισθησία του Sentinel-1 και εδώ βλέπετε ναι. και την ευαισθησία του κόσμου Skymet γιατί τελικά χρησιμοποιήθηκε για έναν εντελώ διαφορετικό σκοπό. Αλλά είναι καλό γιατί τις ικανότητες του δορυφόρου αυτού μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και για έναν άλλο σκοπό που μας βοηθάει στις υποδομές σε μια χώρα όπως είναι η Ιταλία. Και όχι μόνο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρόσβαση στο διάστημα. Η Ιταλία έχει μεγάλη παράδοση. Φτιάχνει εκτοξευτές όπως το Βέγγα που είναι μέρος της οικογένειας εκτοξευτών με το Άριαν 5 και προσεχώς Άριαν 6. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν κάνουμε μεγάλη προσπάθεια από την οποία θα υποφελθεί και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία γιατί συμμετέχει σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά, αλλά συγχρόνως προσφέρουμε και πραγματογνωμοσύνη για τις εξελίξεις των ε, πυράβλων, των μηχανών και οικολογικά. Μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία και όλα αυτά θα τα ξέρει και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει και εκείνη ανάλογα να καθορίσει την πολιτική πρόσβαση στο διάστημα. Αυτά είναι παραδείγματα λοιπόν. Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι άπαξ αυτή η οικογένεια πυράβλων που είναι ανταγωνιστική στο διάστημα μπορεί και οικονομικά να προσφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι θεσμικοί εκτοξευτές να οργανωθούν και να πουληθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υποφεληθεί η αγορά μας χωρίς να καταστραφεί η ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό θέλουμε να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα γίνει αυτό. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και να πώς μια χώρα μπορεί να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Διαστημική ε, Υπηρεσία ώστε να εκπονήσει πολιτικές στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πάμε στις ε, ερωτήσεις, πάμε στις παρατηρήσεις. Ο κύριος Μαρινέσκου εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις έχω. Είναι καλό που η Κορέα χρησιμοποιεί, ακολουθεί το παράδειγμα μας για το έγνος. Το έγνος θα καλύψει όλη τη νέα, τα νέα εδάφη. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε πρόσβαση. Τι σκέφτεστε για τα ποσά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα, τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για το διάστημα από το Brexit και πώς επηρεάζουν και τα αποτελέσματα των εκλογών στις πολιτείες στην κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όσον αφορά την παρατήρηση του ουρανού και του διαστήματος. Σε ευχαριστώ, Μάριαν. Σύντομος και σαφής. Υπέροχα. Ο κύριος Ζανονάτο που εκπροσωπεί τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Σύντομες και σαφείς ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν τελευταίες δύο επιτρέπουν εξίσου σύντομες απαντήσεις, εξίσου σαφείς. Διότι ήταν πολύ γενικού ύφους οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ τους ομιλητές, διότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσίασαν. Τους ευχαριστώ διότι μας έδειξαν και πολύ σαφείς εικόνες της διαφάνειας. Εκμεταλλεύουν ευκαιρία για κάποιες ερωτήσεις, για να διευκρινίσω κάποια σημεία. Το πρώτο ερώτημα. Υπάρχει μεγάλη διεθνής εμπειρία και θεωρώ ότι τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής που παρουσιάστηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να επιτρέψουν στην Ευρώπη να ανταγωνιστεί πραγματικά στο διεθνές πλαίσιο. Μπορούν να επιτρέψουν να ακολουθήσει η Ευρώπη τις εξελίξεις στο διάστημα και στην παγκόσμια αγορά. Πώς αξιολογείται τη θέση μας εν συγκρίση με τον υπόλοιπο κόσμο και με αυτούς που έχουν διαστημική στρατηγική. Δεύτερον, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ίδια ποιότητα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού με όλες τις ε, διεθνείς διαστημικές δυνάμεις. Και πώς μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Κάτι που συνδέεται με την πρώτη ερώτηση. υπάρχουν προβλήματα με τα απόβλητα τα διαστημικά και με τη χρήση ε, λογισμικών και θέματα κυβερνοχώρου όσον αφορά το διάστημα. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε ε, αυτά τα προβλήματα. Προς τον καθηγητή Ματιστών έχω δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά την Ιταλία. Διότι γνωρίζει κάποιες στοιχείες που με απασχολούν. Πρώτον, πώς η Κίνα και η Ινδία αναπτύσσουν δραστηριότητε στο διάστημα και πώς με τις δραστηριότητες τους αλλάζουν την ισορροπία της γεωπολιτικής στο διαστημικό χώρο. Δεύτερη ερώτηση αφορά τη χώρα μου, την κυβέρνησή μου. Ποιε δράσει έκανε η Ιταλία για ενισχύσει τη συμμετοχή την εθνική στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το διάστημα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Αυτά και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κάτω από το χρονικό όριο, υπέροχα και εξίσου σαφής όπως και ο κύριος Μαρινέσκου. Έχουμε υπέροχο αποτέλεσμα. Η κυρία Βανμπόσιουτ εκπροσωπεί το ECR. Πράγματι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές μας για τα ενδιαφέροντα που μας είπαν, για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Μιλώ εκ μέρους συναδέλφου του κ. Σενόφσκι που έπρεπε να αποχωρήσει προς ε, Πράγα. Μου ζήτησε να θέσω δύο ερωτήσεις. Σχετίζονται κάπως με αυτά που ρώτησε ο κ. Μαρινέσκου. Ένα τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GNSS είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση των διαφόρων ε, τσιπ που του Γαλιλαίου υπάρχουν και μηχανισμοί που τα χειρίζονται το GSA. Αρκεί αυτή η προσέγγιση. Δεύτερη ερώτηση. Μελλοντική Βρετανική συμμετοχή στο Γαλιλαίος. το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να είναι ισχυρό στρατηγικός εταίρος. Θα έχει αντίκτυπο το Brexit όσον αφορά το έργο του οργανισμού και κυρίως όσον αφορά το κέντρο ασφαλείας και τις χερσές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπερπόντιες, στα υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασίλειου. Υπέροχα, κυρία μου, διότι υπήρξατε ακριβέστατοι και συντομότατοι. Ε, ανακάλυψε βέβαια ο ίδιος. Ο κύριος Κόχλιτσεκ. Να δούμε αυτός πώς θα τα πάει. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομος, όπως και οι προλαλήσαντες. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτη. Η χρήση, η παρούσα της τεχνολογίας της δορυφορικής για το e-call, κάτι που το συζητήσαμε. Πότε θα εφαρμοστεί. Μετά. Όσον αφορά τα διαστημικά προγράμματα, σε σχέση με τα διαστημικά προγράμματα για τη Ρωσία και την Κίνα, τα προγράμματα αυτών των χωρών, πώς μας επηρεάζουν. Και πώς, πώς, ποια τμήματα των πυράβλων και των εκτοξευτήρων μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκ νέου, να ανακυκλώνεται η χρήση τους. Ήσασταν πάρα πολύ λακωνικός, οπότε να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις και, να, και ίσως να μακρηγορήσω λίγο. Στον πρώτο μιλητή. Πόρη για τον οργανισμό. Στελέχωσης επίσης. Πείτε μας κάτι γι' αυτά. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην ασφάλεια. Τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, Φερρυπίν. Τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Γνωρίζοντα ότι το Γαλιλαίο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή να εκπνεύσει η λειτουργία, μην μπορεί να λειτουργήσει πλέον στο εγγύς μέλλον. Πώς μπορούμε να λειτουργησει πλεον στο εγγυ μελλον πως μπορουμε να κοινοποιησουμε τα ωφέλη του διαστήματος στους λαούς μας. Κάποιος συνάδελφος χτες, παρουσία του κυρίου Σεύκοβιτς και της κυρίας Μπιανκόφσκα το έθεσαν αυτό. Οι φορείς που εκπροσωπείτε, πώς το βλέπουν αυτό. Ο κύριος Μπατιστών τώρα, έχω μια ερώτηση για σας. Είναι περίπλοκη, το, περίπλοκο το σκηνικό το ευρωπαϊκό σαν αυτό το διάστημα. Πώς μπορεί να πλουστευτεί, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ακόμα και για μας να ξεκαθαρίσει εικόνα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στην επόμενη συνεδρίαση της Ίτρε τέλος Νοεμβρίου. Θα τεθεί επισήμω σχετικό ερώτημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα για μας. Τέλος, αλλάζει πρόσβαση στο διάστημα γρήγορα μέσω και ιδιωτικών εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον της ευρωπαϊκής πρόσβασης στο διάστημα. Ίσως να μην υπάρχει αρκετός χώρος στο διάστημα. άλλος της αγορεύειν βούλετε ουδείς. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου συνεχίζει, δυστυχώς δεν ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω απαντώντας τις ερωτήσεις. Από τον κύριο Μαρινέσκου πρώτα. Για την κάλυψη του έγκνος ετοιμάζουμε νέα έκδοση. Θα βελτιωθεί η κάλυψη. Θα καλύπτονται και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποια κενά προς τη Μεσόγειο και Βορειοανατολική Ευρώπη. Για να έχουμε πλήρη κάλυψη πρέπει να πάμε εκτός Ευρώπης και να θέσουμε σταθμό στη Βόρεια Αφρική δεν είναι και τόσο εύκολο πάντα. Ας το θέσω έτσι. Για τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα αρκούν. Να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, να το περιορίσω μάλλον το ερώτημα στο GNSS. Όσον αφορά το GNSS, ο προπολογισμό που διατίθεται σε αυτό το στάδιο ε, θεωρείται αρκετός αλλά όσον αφορά τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει όλη η δυνατότητα να υπάρξει, διότι θα έχουμε σύστημα νέας γενιάς και χρειάζονται χρήματα για την ανάπτυξη αυτού. για τα δύο δύσκολα τελευταία ερωτήματα, το Brexit και τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών. Το Brexit ετέθη και από την κυρία Βαν Μπονσουίτ. Για το Brexit λοιπόν. Να σας πω ότι η Γενική Διεύθυνση Grow είπε να μην προδικάζουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν σύντομα. Ανήκουμε σε μια ομάδα κρούσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αναλύσει ενδεχόμενα προβλήματα. Σε αυτή τη φάση δεν κάνουμε κανένα βήμα. Περιμένουμε. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να διαφυλάξουμε το προσωπικό που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάνω ό,τι μπορώ για να τους κρατήσω τους ανθρώπους αυτούς και είναι πρόβλημα. Για τις πρόσφατες εκλογές τώρα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω. Δύσκολη ερώτηση. Όμως, να σας πω κάτι. Η σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, κάτι σημαντικό, προκαιρού ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Ουάσιγκτον συνάντησα κάποιον αξιωματούχο που μου είπε «Κάρλο, ίσως πριν από δέκα χρόνια να κάναμε λάθος, να είμαστε αντίθετοι με το Γαλιλαίο, αναγνωρίζουμε την αξία που έχει το σύστημα». Και εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούλιο φέτος να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη Δευτέρα θα γίνουν οι πρώτες διαπραγματεύσεις στην Πράγα. Αυτό δείχνει στην Ευρώπη ότι η επιλογή που έγινε πριν κάποια χρόνια ήταν η σωστή. Το ερώτημα του κυρίου Ζανανάτο, αν οι τέσσερι πυλώνες της διαστημικής στρατηγικής είναι αρκετοί για να ανταγωνιστούμε στη διεθνή αγορά. Πιστεύω ναι το έγγραφο, η κοινή δήλωση με τον κύριο Μπατιστόν είναι ένα καλό έγγραφο, είναι περιεκτικό, συνοπτικό, ακριβές, φιλόδοξο, πρέπει να μεταφραστεί και σε συγκεκριμένα βήματα που θα υλοποιηθούν. Μπορούμε να βρούμε εκεί στοιχεία για να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή ε, στο διάστημα και στην παγκόσμια αγορά του διαστήματος. Η άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας εν συγκρίση με τις άλλες ισχυρές διαστημικές δυνάμεις. Και στις διαφάνειες του κυρίου Μπατιστών το είδαμε ότι η Ευρώπη υποφέρει από κατακαιρματισμό ποικιλομορφία κατακαιρματισμού υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, πρώτα απ' όλα, αλλά επιτρέψτε μου να πω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι. Παρεμβαίνουν πολλές γενικές διευθύνσεις. Η μία γενική διεύθυνση δεν γνωρίζει πάντα τι πράττει η άλλη πρέπει να κάνουμε κάτι το ώστε να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση των ωφελημάτων που μπορεί να απορρεύσουν από το διάστημα σιδηρόδρομοι, θαλάσσιες μεταφορές κλπ. Κάτι μπορούμε να κάνουμε εκεί για να διασυνδέσουμε τους διάφορους φορείς και τομείς. Άλλη ερώτηση. Και ο Ζανονάτο για την ε, ασφάλεια αν υπάρχουν προβλήματα. Και ο κύριος Μπιούζεκ ε, παρόμοια ερώτηση έθεσα περί ασφαλείας. Ναι, εστιαστώ επί του GNSS. Είναι ευρύτερη η ερώτηση που το διάστημα. Το GNSS μιλάμε πάντα για ασφάλεια και κινδύνους. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορούμε να εξαλείψουμε τα προβλήματα. Είναι πάντα θέμα υπολοιπωμένου κινδύνου. Έχει σχεδιαστεί το σύστημα αρκετά καλά, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Ποιο είναι το πρόβλημα. Η απειλή κατά της ασφάλειας δεν είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι που αλλάζει. Δεν θα έλεγα καθημερινά, σχεδόν όμως. Ποια είναι η δυσκολία αντιμετωπίζουμε νέες απειλές και να παρακολουθούμε τι γίνεται εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που διαβλέπω. Να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά το GNSS δίδεται μεγάλη προσοχή. Και μπορούμε να πούμε ότι εν γέννη καλά τα πάμε. Το ερώτημα της κυρίας Βαν Μποσούιτ για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για το Γαλιλαίος και τα τσιπάκια. Μας είπαν πρόσφατα κάποια καλά πράγματα, καλά μαντάτα. Γι' αυτό έχουμε 40% μοντέλων και συσκευών που έχουν προγραμματιστεί να λειτουργούν με το Γαλιλαίος. Είναι καλά μαντάτα, διότι το σύστημα δεν είναι πλήρως λειτουργικό είναι αποτέλεσμα μεγάλων προσπαθειών που έκανε ο οργανισμός συνομιλώντας πολύ συχνά σχεδόν εβδομαδία με τους αρμόδιους φορείς όλο τον κόσμο. Με τους Αμερικανούς, με τους Ασιάτες. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές προσπάθειες που κατεβλήθησαν στην Ευρώπη. Έχουμε ένα φορέα στην Ευρώπη μόνο που συμμετέχει σε Εδώ ίσως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Βασικό στοιχείο, και σωστά το αναφέρετε, είναι τα χρήματα. Αποκλειστική πόρη για να αναπτύξουμε τους δέκτες για το GNSS είναι 100 εκατομμύρια για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αρκεί ποτέ δεν αρκετά τα χρήματα. Εν γέννη δεν επενδύουμε πολλά στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών και δεκτών ε, για το Γαλιλαίος. Ε, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και αυτό ε, στις επόμενες δημοσιονομικές πλωτικές και αυτό εν συγκρίση πάντα με το τι κάνουν οι ΙΠΑ. Αυτά σε σχέση με το Brexit. Τώρα για τους πόρους. Ερώτηση του κ. Μπούζεκ. Έλεγα ουσιαστικά 103 είμαστε φέτος, αν δείτε τη διάσταση, τις επενδύσεις που χειριζόμαστε, τις πολλές κατευθύνσεις στις οποίες κινούμεθα, μπορώ να σας πω ότι είναι πρόβλημα καθημερινό να εργαζόμαστε σωστά. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι βασιζόμαστε κατά πολύ σε υπεργολαβίες, σε αναθέσεις, σε φορείς ε, παροχή συμβουλών και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Και στο τέλος της... των συμβάσεων έχουμε προβλήματα. Εγώ σχεδιάζω σύντομα να παρουσιάσω νέο αίτημα για κονδύλια στην Γενική Διεύθυνση Growth για να πετύχουμε καλύτερη ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ φόρτου εργασίας, ευθυνών και πόρων για την επικοινωνία κλπ. Πολύ σωστό αυτό. Πάντα υπάρχει πρόβλημα εδώ. Χρειάζεται να προβάλλουμε την εικόνα μας, να επικοινωνούμε με τα διάφορα ακροατήρια, να δείχνουμε τα ωφέλη που αποκομίζει η χρήση του διαστήματος και του στήματος του δορυφορικού Γαλιλαίος. Το πρόσφατο παράδειγμα θα είδατε το θόλο που είχαμε εδώ στις Βρυξέλλες αυτός ο θόλος έδειχνε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με το σύστημα Γαλιλαίος αλλά και αλλού. Ταξίδευε αυτός ο θόλος όλη την Ευρώπη και φτάσαμε τους ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι ένα καλό παράδειγμα. Δείχνουν πώς μπορούμε να ε, μαζευτούμε όλοι μαζί και να κοινοποιούμε με καλύτερο τρόπο στο κοινό τα ωφέλη του διαστήματος. Ευχαριστώ και ως Μπατιστών, ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν. Κάποιες από αυτές ήδη καλύφθηκαν από τον κύριο Ντεντορίντ. προπολογισμό. Δείχνουν αναλύσεις ότι η επένδυση στο διάστημα πολλαπλασιάζει την επένδυση από δύο, μέχρι, δύο φορές μέχρι 6-7 φορές την αρχική επένδυση. Από, την πολλαπλασιάζει. Είναι σωστή η ανάλυση. Αυτή έχει γίνει σε διάφορα περιβάλλοντα, σε διάφορες χώρες. Είναι σίγουρο αυτό ότι πολλαπλασιάζει την επένδυση στο διάστημα. Η επένδυση στο διάστημα είναι επικερδής, αξίζει τον κόπο, ωφελεί την οικονομία και την κοινωνία η διαφάνεια και ο χάρτη σα, το, το πίνακα σας έδειξα, έδειχνε ότι η Ευρώπη αποτελείται 500 περίπου εκατομμύρια ανθρώπου είναι πιο μεγάλη από τη ΣΥΠΑ σε πληθυσμό και τη Ρωσία, θα μπορούσαμε να είχαν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις για το διάστημα. Ο ουρανός είναι το όριό μα όπω είπε εδώ. Χρειαζόμαστε επενδύσει επένδυση το διάστημα. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και με τι άλλε δραστηριότητε, αλλά το διάστημα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, προωθεί την οικονομία, άρα αποτελεί κινητήρα για αναζωγόνηση και πρόθεση της οικονομίας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι όσον αφορά αυτό. Δεν υπάρχει κάτι μαζικό που μπορούμε να κάνουμε με τον προϋπολογισμό που, έχουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία δεκαετία έχει παρεμβαίνει και έχει αλλάξει την εικόνα του διαστήματος, η παρέμβασή τη, αλλά ακόμα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ τώρα. Από τη ΣΥΠΑ ήρθα τώρα. Εκεί την περίφημη νύχτα ήμουν εκεί. Δάκρυσα, βούρκωσα, τι να σας πω. Ψηφίσατε, ρωτάει και ο Σμπούζεκ. Όχι βέβαια. Πολύ παράξενη νύχτα, ιδιαίτερη. Το σκεφτόμουν επιστρέφοντας. Τα πράγματα θα αλλάξουν, σίγουρα. Ίσως λιγότερο από ό,τι περιμένουμε, θα αλλάξουν. Ένα είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας σε κάποιους τομείς. Ακόμα και σε, κάποιες, σε κάποιους χώρους του διαστήματος. Κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά. Αυτό είναι πρόκληση αλλά και ευκαιρία για το SST, το PRS, για το Γαλιλαίος. Είμαστε μόνοι μας. Πρέπει μόνοι μας να κινηθούμε προς το μέλλον. Να είμαστε θετικοί όμως στην προσέγγιση. Να μην βλέπουμε όλα αυτά μαύρα και δυσκολίες. Αυτά που έθεσε ο κύριος Ζανονάτο, τα σχόλιά του. Αν οι πυλώνες του όλου εγχειρήματο για τη διαστημική στρατηγική, αν είναι σωστή, οι προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση στρατηγικής και τη σύνταξη του εγγράφου ήταν όλα καλά. Τα χαιρετίζουμε. Σαν Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε συναντώμενοι και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες φορές. Ναι, είναι καλή αφετηρία, εξοχή αφετηρία θα έλεγα, αλλά πρέπει να δούμε ότι είναι πολύ νέο τομέα το διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 40 ετών. Ξεκίνησε στη Λισαβόνα την τελευταία δεκαετία η υλοποίηση. Έχουμε τεράστια πρόοδο εν μεταξύ, συγγνώμη, και καταλήξαμε σε πολλά αποτελέσματα. Αυτό είναι καλό έγγραφο, αντικατοπτρίζει αρκετά καλά την παρούσα κατάσταση σε δύο-τρία χρόνια πρέπει να προβούμε σε μια αναθεώρηση, διότι αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά καλή αρχή. Μεταξύ πολλών που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν τα χρήματα. Τα χρήματα μια πολιτική απόφαση μπορεί να διατεθούν, δεν είναι τεχνολογία, διότι η Ευρώπη έχει έξοχη τεχνολογία σε πολλούς τομείς, εξαιρετικές βιομηχανίες, διανεμημένες σε διάφορες χώρες. Το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο. Η νοοτροπία που φοβάται το κίνδυνο με προβληματίζει. Είναι η νοοτροπία της Υπήρου όσον αφορά τις επενδύσεις. Και τα διάφορα παρεπόμενα ωφέλη και προϊόντα. Δηλαδή υπάρχει νοοτροπία ότι αν αποτύχει κανείς ε, είναι νεκρός, ενώ από την άλλη μεριά Ακόμα και αν αποτύχει πολλέ φορέ, θα πετύχει τελικά. Το ξανακάνει, το ξανακάνει μέχρι να πετύχει, λένε οι Αμερικανοί. Και μάλλον είναι και καλό χαρακτηριστικό στο βιογραφικό για του Αμερικανού αν αποτύχει κανεί και τελικά πετύχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πιο δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει μέσω απόφαση, ε, μέσω εγγράφου κλπ. Είναι θέμα πολιτισμικό η επένδυση. Ίσως στην Ευρώπη οι διάφορες χώρες μπορεί να συμβάλλουν με διαφορετικές νοοτροπίες. Αυτό είναι ο πλούτος. Έχουμε διαφορετικούς ε, πολιτισμούς και νοοτροπίες που εμπλουτίζουν τη γενικότερη νοοτροπία. Αλλά αυτό όσον αφορά το διάστημα είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Να μπορεί κανείς να αρπάξει την ευκαιρία που δίνει το διάστημα που αλλάζει γρήγορα και να αναλάβει τον κίνδυνο και να είναι φιλόδοξος. Κίνα και Ινδία. Αυτά αφορά την ισχύ τη υγεία, ε, συγγνώμη, ε, τεχνολογίας και της επιστήμης που διαμορφώνει την ε, διπλωματία στο διάστημα. Και είναι πολύ ισχυρό εργαλείο η διαστημική διπλωματία. Δημιουργεί και δεσμούς. Ξεπερνάει τείχους, δύσκολες εποχές και βοηθά τη συνεργασία. Έχω 20 χρόνια εμπειρία συνεργασίας με την Κίνα. Ας συνεργαστούμε όσον αφορά την εξερεύνηση, να πάμε στο, στη Σελήνη, στον Άρη με αυτές τις χώρες, στην επιστημονική έρευνα κλπ. Διότι έτσι θα ανοίξει ο χώρος ο οικονομικός, ο βιομηχανικός και ο πολιτικός. Που πιο εύκολα να ξεκινήσουμε από εκεί από ό,τι στους άλλους χώρους που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε πολλά για να ενισχύσουμε τη συνεργασία στο διάστημα για την Ιταλία. Το απάντησα. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να ακολουθήσουμε πιο σφαιρική και συντονισμένη προσέγγιση. Και καλά πηγαίνει αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια τα κονδύλια για, την, ε, για, την οργαν, τον οργανισμό μας αυξήθηκαν. Διετέθησαν νέο πόροι φέτος το καλοκαίρι για την Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος και έτσι τονώνεται και η οικονομία και η συνεργασία εταιριών με το δημόσιο τομέα. Μετά, Θέσατε ερωτήσει και εσείς κύριε Πρόεδρε. Η εικόνα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διάστημα είναι περίπλοκη. Έχω ένα σχόλιο. Πριν τη Λισαβόνα, τη συνθήκη τη Λισαβόνα, πριν μπει στο παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα. είχαμε εθνικού οργανισμού και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο και όλα λειτουργούσαν αθόρυβα. Ήταν σαφή ο ρόλο τη ΕΖΑ, των εθνικών επίσης φορέων, σαφής ο ρόλος, και ίδρυσαν οι εθνικοί φορείς στην ΕΖΑ, ούτω ώστε να συναθρίζονται αρκετοί πόροι για να μπορούμε να κατασκευάζουμε πυράβλους που μπορούμε να μεταφέρουν μεγάλα φορτία, να ανακαλύψουμε το σύμπαν, να αναπτύξουμε τεχνολογίες για επικοινωνίες, για ε, ανείχνευση της γης κλπ. Κάτι που δεν μπορούσε ένας εθνικός φορέας να κάνει μόνος του από όταν μπήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ φιλόδοξες και σημαντικές στρατηγικές, από τότε έχουμε υπολείμματα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο αυτών φορέων. Και αν δεν κάνουμε κάποια βήματα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ποιος κάνει τι, ούτω ώστε η ΕΖΑ να μην φοβάται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υποτιμά την ΕΖΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο θα έχουμε συνεχώ δυσκολίε. Είμαι πολύ νέο στον τομέα. Μόνο δυόμιση χρόνια είμαι εδώ. Δεν μπορώ. Μπορεί να δίνω κάποια νέα άποψη. Σωστή ή λάθο. Αυτό αισθάνομαι όμω. Αυτό σας λέω. Ήρθανε κάποιοι νέοι φορείς, πολύ μεγάλος, σημαντικός νέο φορέας μπήκε άλλαξε ισορροπία και δεν είναι σαφή ικανότητα του παιχνιδιού. Αν κάνουμε προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν αυτοί, η ΕΣΑ έχει τεράστιε δυνατότητε. Είναι το σύνολο τη τεχνολογία, τη γνώση, τη εξερεύνηση των νέων πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Πίεση Διαστήματο. Και να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει του μεγάλου στόχου μέσω τη τεχνογνωσία που έχει η ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τα κοινωνικά ωφέλη κλπ και άλλη την τεχνολογία. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τα όρια μεταξύ των δύο πλευρών και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί, αυτή η θολούρα δημιουργεί προβλήματα. Ερώτηση του κ. Μπούζακα. Επιτρέψτε να σα ρωτήσω. ΕΖΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι. Η GSA, που είναι εδώ δίπλα μας. Ναι, πολύ καλή ερώτηση που λέει Η GSA είναι η προσπάθεια που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλάβει ικανότητε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δεν βλέπω τίποτε κακό σε αυτό. Γιατί είναι ευρωπαϊκές υποδομές ο Γαλιλαίο. Και μπορεί να είναι ή όχι το σώμα το οποίο θα τον τρέξει, θα τον φέρει σε λειτουργία. Απόλυτα θεμητό να αναλάβει την διαχείρισή του μια ευρωπαϊκή υπηρεσία. Μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο και κόπο, αλλά δεν το βλέπω κακό, γιατί η ΕΖΑ, μακροπρόθεσμα ίσως, ε, ανταγωνίζεται για να λάβει τη σχετική αρμοδιότητα. Δηλαδή, όμως μας λέτε ότι είναι ρυθμιστικό σώμα η GSA. Όπως και η Επιτροπή δηλαδή. Από τη θεώρηση της ε, ρύθμισης, ναι, Αλλά εμείς εστιάζουμε στην λειτουργία και την παροχή υπηρεσίας. Επομένως, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη, σε δική μας περίπτωση, του συστήματος. Επομένως, παίρνουμε το σύστημα και το εστιάζουμε στην, παρεχ... στην προσπαροχή υπηρεσία. Σε αυτό δεν έχουμε ανταγωνιστική σχέση με την ε, ΕΖΑ, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Υπάρχουν κάποια άλλα στα οποία μπορεί να υπάρχουν ε, άλλες αξιολογήσεις πριν από μερικά χρόνια, όπου είχαμε την ε, παραγωγή προϊόντος από την ΕΖΑ που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι σε ανταγωνιστική σχέση με εμάς. Δηλαδή ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συστήματος δεν είναι ρυθμιστικό σώμα, έτσι. Δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Ναι, έχει σημαντικό ρόλο στην ε, διαμόρφωση βιομηχανικής πολιτικής, αλλά δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Και αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμη, ένα σχόλιο για την πρόσβαση στην αγορά και κάτι που αναφέρατε κι εσείς. Συγκεκριμένες ιδέες. Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς ως κερδοφόρο ε, δραστηριότητα την εκτόξευση πυράβλου. Είναι πολύ περισσότερο το κόστος, είναι πολύ περισσότερη η πύραυλη που έχουμε εμείς εκτοξεύσει από ό,τι θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει από κάποιον αντίστοιχο φορέα στον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Μέσα σε 100 χρόνια μπορεί να υπάρξει κάποια σχέση οικονομία κλίμακας, αλλά όχι τώρα. Όπως λειτουργεί η οικονομία, χρειάζεται ούτω ή άλλω δημόσια επένδυση. Με τη μεγαλύτερη πρόκληση στο SpaceX. Δύο διαφορετικές τιμές προσφέρει στην NASA και την AOD για την κάλυψη των ε, αναγκών σε υπηρεσίες των μεγάλων πελατών. Εδώ στην Ευρώπη, με την Υπουργική 2014, κάναμε μια τεράστια, ένα τεράστιο άλμα με την ΕΖΑ, στη συνεργασία με τον κλάδο. Να καλύπτει ο κλάδος της ανάγκης και όχι η ΕΖΑ μεγάλο άλμα, σημείο καμπής, αλλά έχει τεράστια σημασία. Και από εδώ και μπρος, από το 2020 συγκεκριμένα, ο κλάδος ο οποίος έχει την δραστηριότητα της εκτόξευσης είναι πια μόνος του, χωρίς την υποστήριξή μας και βεβαίως έχει σε μεγάλο βαθμό δράση εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μεγάλος πελάτης. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν το ερώτημα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σεβασμού προ το δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτόνομη παρουσία στο διάστημα, αλλά το επιχειρησιακό σχήμα πάνω στο οποίο θα εργαστούμε για να φέρει αποτελέσματα δεν είναι βιώσιμο στη μορφή που έχει τώρα. Θα καταρρεύσει. Α μην κρυβόμαστε. Κανείς, Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Κίνα, η πιο ε, εύπορη καπιταλιστική βιομηχανική ε, επιχείρηση δεν μπορεί μόνη της να σταθεί. Το αποκλείω. Κύριε Κόβιτσικ, ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ζητώ συγγνώμη σας να μην έγιναν κατανοητή η ερώτησή μου. Ναι. Αν θέλετε να σας την επαναλάβω στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τι προτιμάτε. Χρήση οίκορ από, τις, ε, από τους πυράβλους. Και δεύτερον, πόσοι είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιεί το σύστημα Γαλιλαίος στο διάστημα. Τρίτον, πρόγραμμα COSMIC και σχέση της υπηρεσίας σας με τη Ρωσία και την Κίνα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Και η έννοια της επαναχρησιμοποίησης των, εκπυρσο... των ε, για τους ε, πυράβλους, των εκτοξευτών, ναι, ευχαριστούμε και πάλι. Βέβαια δεν ήταν ε, σωστό ότι επαναλάβατε, είχατε την ευκαιρία να επαναλάβετε. Αν θέλετε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και την επόμενη ομάδα. Ναι, βεβαίω, πολύ σύντομα και ζητώ συγγνώμη που δεν έδωσε επαρκή απαντήσει στην ερώτησή σα. Δεν δουλεύουν καλά τα ακουστικά μου, φαίνεται. Λοιπόν, από το 2018 όλα τα αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εξοπλισμένα με το σύστημα Γαλιλαίος. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι είμαστε σε ε, εντατικέ συνομιλίες με την αυτοκινητοβιομηχανία και αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να παρημπρώσει η βιομηχανία, η αγορά σε σχέση με τον Γαλιλαίο και να τον ενσωματώσει. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η χρονολογία το 2018. Πόσους δορυφόρους έχουμε στο διάστημα. 14 αυτή τη στιγμή. Την επόμενη εβδομάδα, 17 του μηνός, θα έχουμε την πρώτη εκτόξευση από τη Γαλλική Γουιάννα τεσσάρων ταυτόχρονα δορυφόρων. Πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Έτσι θα είναι συνολικά μέχρι το τέλος του 16-18 του χρόνου άλλο ένα, άλλη μια εκτόξευση αριάν 5, δηλαδή άλλους 4. Ευχαριστώ που επαναλάβατε την ερώτηση. Η συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα. Έχουμε με την Κίνα επιστημονική συνεργασία σε δύο τομείς. συλλογή δεδομένων καταρχάς από, τα, από ένα από τα δύο κινέζικα παρατηρητήρια και παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης της επιφάνειας της σελήνης με πληροφορία πολλαπλού φάσματος, ώστε να είναι διαθέσιμες πληροφορίες στην καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και επίσης παρατήρηση ε, φαινομένων από το διάστημα που μπορεί να έχουν σχέση με γεωφυσικά φαινόμενα, θερυπίν ε, σεισμοί. Τους παρατηρούμε από το διάστημα και σε αυτό έχουμε αναπτύξει τέτοια διπλωματία του διαστήματος με την Κίνα και θέλουμε να την ε, επεκτείνουμε περαιτέρω, να βρούμε τρόπους συνεργασίας και έχουμε συμμετάσχει και στην ανάπτυξη του επανδρομένου δορυφορικού σταθμού της Κίνας που μπορεί να έχει πολύ σημαντική χρησιμότητα για τη χώρα αυτή. Ρωσία. Συζητούμε εφαρμογές σε μελέτες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές. Επεκτείνουμε τις δραστηριότητε μας σε σταθερή, σταθερό στη σημείο σε σχέση με την υγιή ε, σε τροχιά και αυτό πάλι, πάλι στο χώρο της παρακολούθησης των κλιματικών αλλαγών. Επαναχρησιμοποιήσαμε η δεύτερη ερώτηση. Η ΕΖΑ ξεκινάει με μελέτες για την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης με ένα νέο πρόγραμμα που συζήτησε και η Υπουργική Συνήθω για ένα μελλοντικό τύπο πυράβλου θα έλεγα θα ήταν ο Αριάν 7. Σε αυτό τίνουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο και τους δύο ομιλητέ, εξαιρετικέ οι ε, ομιλίε τους, όπω και οι απαντήσει, τους, πολύ ενδιαφέρουσε. Και τώρα περνώ στο δεύτερο πάνελ και τον κύριο Τόρτορα και τον κύριο Προύναριο τους οποίου και καλό να έρθουν στο Προεδρείο. Ο κύριος Τόρτορα, πρώτος, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτικής για το Διάστημα. Δεν είναι ακόμη η υπηρεσία. Την επόμενη φορά θα έχει μετατραπεί σε υπηρεσία στην επόμενη μας συνεδρία. Σε Ευρωπαϊκό λοιπόν Ινστιτούτο Πολιτικής για το Διάστημα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρόκειται για έρευνα, επιστημονική πάντα, τεχνική φύσεως ίσως, Έρευνα βάσης επίσης. Έχετε να μας πείτε τίποτα για όποια καινοτομία έχετε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουζεκ. Ευχαριστώ πολύ που με καλήσατε εδώ να έρθω να μιλήσω για τη νέα μου θέση πριν από ένα μήνα περίπου ανέλαβα. Οπότε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικής ε, Πολιτικής είναι ένα think tank που αφοσιώνεται σε προβληματισμό και μελέτες όσον αφορά τις επιθυμητές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική. Εξετάζει βέβαια και το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Η έδρα είναι στη Βιέννη. Πολύ καλό μέρος να βρίσκεται μια τέτοια δραστηριότητα γιατί είναι ένα παράθυρο ανοιχτό προς τον κόσμο, γιατί υπάρχουν εκεί και οι Ηνωμένα Έθνη και άλλοι οργανισμοί όπου γίνονται διεθνείς συζητήσεις όσον αφορά την νομοθεσία του διαστήματος. Αυτά λοιπόν για την αποστολή του Ινστιτούτου μου, το οποίο και εκπρόσωπο εδώ σήμερα μου ζητήσατε να σας μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα. Προηγουμένως όμως θέλω να αρχίσω με ευχαριστίες. Συνήθω στο τέλος της παρουσίασης δίνονται ευχαριστίε. Εγώ θα αρχίσω με τι ευχαριστίες. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτ. ευχαριστώ την Επιτροπό Μπιέκοφσκα, ευχαριστώ την Γενική Διεύθυνση Κρόου, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και τι χώρε μέλη που βάζουν το διάστημα στην κορυφή τη Ευρωπαϊκή πολιτική Ατζέντα για το 2016. Είναι σίγουρα μια πολύ καλή πρωτοβουλία και σίγουρα την κατάλληλη στιγμή συζητούμε για την προβληματική αυτή και ευχαριστώ πολύ και το Πακό Κοινοβούλιο για την στήριξή του γιατί πολλά διακυδεύονται εδώ. Αλλά θα περιοριστώ όπως σας είπα στην ανταγωνιστικότητα τώρα και τα σχετικά. Ανταγωνιστικότητα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Περί πρόκειται όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο ανταγωνιστικότητας, γιατί δεν πρόκειται για μια απόλυτη τιμή, αλλά για μια σχετική τιμή. Είσαστε ανταγωνιστικός σε σύγκριση με κάποιον άλλον. Δεν μπορείτε να, είσαστε, να πείτε ότι είσαστε ανταγωνιστικός μια για πάντα. Όχι. Φτάνετε σε ένα επίπεδο ανταγωνιστικότητας και μετά πρέπει να λάβετε υπόψη σας την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των ε, δυνατοτήτων που έχετε εσείς, αλλά και ανταγωνιστές σας. Αλλού στον κόσμο. Η ανταγωνιστικότητα γι' αυτό πρέπει να βελτιώνεται αδιάκοπα. Είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος. Πρέπει να στηρίζεται για πάντα. Μπορεί να ακούγεται αποθαρρυντικό, αλλά έτσι είναι. Και ακόμα και όταν οι ανταγωνιστές σας δεν κάνουν τίποτα, κάτι το οποίο δεν ισχύει τώρα, άρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια αυτή για ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, μια από τις δυσκολίες που έχουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, είναι να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το δικό μας επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να μπούμε στη διεθνή αγορά και να ανταγωνιστούμε εκεί. Βάσει αυτής της υπόθεσης λοιπόν, σήμερα μπορούμε με αρκετή εμπιστοσύνη να πούμε ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι ανταγωνιστική. Γιατί αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητά της κάθε φορά που έχει την ευκαιρία να δείξει πόσο ανταγωνιστική είναι σε ανοιχτές και σωστές αγορές με συγκεκριμένους στόχους. 43% ουσιαστικά ήταν το μερίδιο του τζίρου στις εμπορικές αγορές το 2015. Η κατάσταση αυτή παγκοσμίω είναι μοναδική. Αλλά κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι η ανταγωνιστικότητα είναι βιομηχανική υπόθεση. Και θα συγκρίνω την κατάσταση με το τι γίνεται στην επιστήμη. Κανείς δεν θα πει ότι η επιστημονική κοινότητα πρέπει να αποφασίσει για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ετοιμαστούν οι επόμενες επιστημονικές ε, αποστολές. Αλλά για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα, πολλοί κόσμος έχει πολλές και διάφορες ιδέες. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά αν θέλετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να βασιστείτε εκτενέστατα στην ίδια την βιομηχανία, στις ανάγκες της και τις προτάσεις της. Και αρνούμε ότι οποιοδήποτε άλλος είναι σε θέση να κάνει σαφή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που πρέπει να αναλάβουμε για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Αν πρόκειται για άλλους στόχους, πέρα της ανταγωνιστικότητας, να ετοιμάσουμε θεσμικές αποστολές κτλ. Εντάξει, αλλά μιλάμε για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και μόνο, τότε είναι η βιομηχανία αυτή η οποία θα θέσει τους στόχους. Στις διαδικασίες που έχουμε σήμερα για την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας των ε, δημοσίων, των κρατικών, των προγραμμάτων έρευνας ε, και ανάπτυξης, η βιομηχανία γνωματεύει μόνο. Έχει συμβουλευτικό ρόλο και τίποτα παραπάνω. Θα έπρεπε να έχει παραπάνω όμως ρόλο. Τώρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για στήριξη της ανταγωνιστικότητας, ούτε και αυτό είναι εύκολο να πούμε τι πρέπει να γίνει. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε δημόσια στήριξη στην ανταγωνιστικότητα. Η απάντησή μου, η σύντομη, είναι γιατί χρειάζεται να έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνιστικότητας με τους ανταγωνιστές μας. Και γιατί δεν έχουμε ισότιμους όρους τώρα? Γιατί δεν υπάρχει ισορροπία στις εσωτερικές αγορές, στις διάφορες περιοχές του κόσμου και σήμερα η ευρωπαϊκή θεσμική ζήτηση είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Ή στη Ρωσία, ή στην Κίνα, την Ιαπωνία ή και αλλού, όπου υπάρχουν διαστημικές δυνάμεις. Όπως είπα, έχουμε 43% τζίρο στις εμπορικές αγορές από το διάστημα. Άρα 57% στις θεσμικές αγορές. Δεν έχει ξανακουστεί αυτό. Στις Ηνωμένε Πολιτείε θα ήταν 80%, στη Ρωσία σχεδόν 100%, στην Κίνα σίγουρα είναι 100%, στην Ινδία επίσης και στην Ιαπωνία επίσης 100%. Συνεπώς, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το γεγονός ότι η ζήτηση στην Ευρώπη είναι διαφορετική από ό,τι μεταξύ των ανταγωνιστών μας. Δεύτερον, περί τίνος πρόκειται. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να ε, διασφαλίσουμε απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους ε, τομείς τεχνολογίας του διαστήματος. Αν μία επιχείρηση δεν είναι σε θέση να προσφέρει έχοντας ε, πρόσβαση σε όλη τη διαστημική τεχνολογία αυτό που ζητάει ο πελάτης, τότε βγαίνει από την αγορά. Άρα είναι θέμα επιβίωσης να υπάρχει αυτή η απεριόριστη πρόσβαση και μάλιστα με λογικές οικονομικές συνθήκες. Και εδώ έρχονται τα προγράμματα δημόσιας εγγύησης. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Όπως είπα και πριν, πρέπει να βασιστούμε στην αξιολόγηση που κάνει ο κλάδος για τις ανάγκες. Προς το παρόν η κατάσταση είναι αρκετά ευνοϊκή, γιατί εγώ δεν ξέρω καμία άλλη περιοχή στον κόσμο όπου ο κλάδος να μπορεί να καθίσει γύρω από το ίδιο τραπέζι και από κοινού να συζητήσει συνενετικά για το χάρτη πορείας που χρειαζόμαστε για τις τεχνολογίες. Και αυτό είναι κάτι από το οποίο πρέπει να αποφεληθούμε. Και βέβαια πρέπει να δούμε τα πράγματα ανατομέα. Να δούμε αν ας πούμε πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα στην ε, παρατήρηση της γης σε σχέση με την πλοήγηση ή όχι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, είναι μια πολιτική απόφαση σε ένα τομέα πάντως ο κλάδος είναι σε θέση να καθορίσει προτεραιότητες. Και δεύτερον, πρέπει να πετύχουμε υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας. Τα προγράμματα εγγύησης σήμερα επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμα προγράμματα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τεχνολογιών, το οποίο είναι πολύ καλό αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα, τότε δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Η ανταγωνιστικότητα έρχεται με υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας. Αυτό και η βιομηχανία χρειάζεται προϊόντα. Όπως είπα, η θεσμική ζήτηση στην Ευρώπη είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας, αν λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος της Ευρώπης. Έπειτα, ανάπτυξη εσωτερικών αγορών για υπηρεσίες που βασίζονται στο διάστημα. Όπως το λέει και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι εφικτά για μη οικονομική στήριξη στην διαστημική βιομηχανία, που είναι ευπρόσδεκτα βέβαια. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Οικονομική Διπλωματία. Και αυτό αναφέρεται στο εγγραφό της Επιτροπής. Καλή πρωτοβουλία. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για το διάστημα, όπως και η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως υπάρχουν και άλλες μη οικονομικές που είναι σημαντικές. Θα σα αναφέρω την προβλεψιμότητα των προπολογισμών, οι μακροπρόθεσμες πολιτικές δεσμεύσεις, η διαφάνεια και σταθερότητα των κανόνων, η ασφάλεια των υποδομών. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των καινοτόμων προγραμμάτων προμήθειας έχουν να κάνουν με την εξέλιξη στη σχέση των ε, θεσμικών παραγόντων με τον κλάδο. Θα επανέλθω σε λίγο. Γιατί το κύριο σημείο είναι ότι για πρώτη φορά στο θέμα των ε, μεταφορών στο διάστημα οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισαν να μετακινηθούν από τη θέση του ε, πελάτη που καθορίζει τις τεχνολογικές προδιαγραφές κτλ. στην ε, θέση του καταναλωτή. Κάτι το οποίο έχει πολλές επιπτώσεις στον κλάδο και στις σχέσεις. Η Ευρώπη λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη να κάνει αυτή την αλλαγή. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Και για να ολοκληρώσω, γιατί έχω εξαντλήσει το χρόνο μου φαντάζομαι, θέλω να αναφερθώ σε μερικά θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στο έγγραφο της Κομισιόν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συζητηθούν γιατί θα απασχολήσουν τις εξελίξεις. Είναι το θέμα της ασφάλειας στο διάστημα πρώτα απ' όλα, γιατί νέο διάστημα σημαίνει και νέες απειλές. Γιατί όλο και περισσότερα αντικείμενα ε, εκτοξεύονται, αλλά και γιατί πολλαπλασιάζονται και οι φορείς. Έπειτα υπάρχει το θέμα του κρυφού εξοπλισμού. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχω ακούσει καμία απολύτω ευρωπαϊκή θέση. Και όμως είναι κάτι που πρέπει να λυθεί υπόψη. Και εδώ θα κάνω έναν παραλληλισμό με το τι γίνεται στο κυβερνοχώρο. Με τους ε, εκτοξευτές, το r και το Vega, είναι πολύ καλά μέσα για να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα τμήματα των αναγκών. Αλλά σήμερα δεν ασχολούμαστε με τους πολύ μικρούς εκτοξευτές για τους πολύ μικρούς δορυφόρους. Ξέρουμε ότι επεκτείνεται πάρα πολύ αγορά. Η Ευρώπη τι θα κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει στα χέρια του ιδιωτικού τομέα ή πρέπει και οι θεσμοί να ασχοληθούν το δημόσιο. Και την άλλη μεριά έχουμε βέβαια και αντίθετα τους πολύ βαρύς εκτοξευτές. Στι Ηνωμένε Πολιτείε φτιάχνεται ένας. Αλλά στο μέλλον, με μια διεθνή συνεργασία για την εξερεύνηση του διαστήματος, θα έπρεπε να έχουμε την ικανότητα για βαρύς εκτοξευτές και υπάρχουν και κάποια άλλα. Ε, η νομοθεσία για το διάστημα. Μια που όπως είπαμε οι διάφοροι φορείς, δημόσιοι, ιδιωτικοί πολλαπλασιάζονται. Είναι το θέμα λοιπόν της κίνησης, της μεταφοράς γύρω από το διάστημα και είναι και το θέμα της ε, διαχείρισης, διακυβέρνησης του διαστήματος. Και τέλος, το τελευταίο μου είναι ακριβώς η εξερεύνηση του διαστήματος. Σήμερα δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις και ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Ευρώπης από αυτού. Γίνονται πολλές συζητήσεις στη διεθνή σκηνή και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να συμμετέχει και η Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Προυμαρίου, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρουμανικής Διαστημικής Υπηρεσίας και κοσμοναύτης, αστροναύτης, ε, τώρα ή τέος. Πριν από 35 χρόνια. Ε, έπρεπε να σας ρωτήσω όμως. Μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τα όσα θα μας πείτε, να ακούσουμε αυτά θα μας πείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διεκεκριμένο κρατήριο κύριε Πρόεδρε. Είμαι κατοστός άνθρωπος του πλανήτη που είδε την ομορφιά του πλανήτη από το διάστημα. Είναι μοναδικό ο πλανήτης Γη, αν τον δει κανεί από ψηλά δεν βλέπει κανεί σύνορα, δεν βλέπει συμφέροντα, δεν βλέπει δολοπλοκίε και δεν βλέπει κρίσεις. Βλέπει κανείς ε, ότι είναι έθρωτο και ευάλωτο. Είναι πολύ λεπτή η ατμόσφαιρα, μα συγκλονίζει. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ λεπτή που εξασφαλίζει τη ζωή στην Γη ε, διότι ε, υπάρχει άγνοια εκείνων που ρηπαίνουν την γη, και έτσι ε, μειώνουν τους πράσινους ε, πνεύμονες της γης που μας δίνουν το αναπνεύσιμο οξυγόνο και δεν καταλαβαίνουν ότι υπονομεύουν την υγεία και την ύπαρξη μελλοντικών γενιών. Έχοντας την εμπειρία του διαστήματος και έχοντας ε, ψηλέ θέσεις σε διάφορου οργανισμούς στη γη, γνωρίζω σε ποιο βαθμό η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ζωτική σημασία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η προθυμία και η διεθνή συνεργασία και έχω μεγαλύτερη επίγνωση του τι εμείς ε, το ανθρώπινα όντα μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε και να επενδύσουμε στην επένδυσή μας για το μέλλον, τις αξίες μας σαν ανθρωπινό είδος, σαν ένωση, σαν κράτη. Σημαντικά πρόσφατα σαν μέλος μιας task force εντός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Στατηγικών Μελετών στην ανάπτυξη μιας μελέτης όσον αφορά την ασφάλεια του διαστήματος για την Ευρώπη. Θα χρησιμοποιήσω κάποιες σκέψεις από αυτή τη μελέτη, σε αυτή την παρουσίαση. Περίπου 1.300 δορυφόροι είναι γύρω από τη γη, ε, ανήκουν σε πάνω από 8 χώρες και οργανισμούς και παρέχουν ε, πλήθος πληροφοριών για δισεκατομμύρια ε, ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 18 δορυφόρους που είναι σε τροχιά και έχει προγραμματίσει πάνω από 30 για τα επόμενα 10-15 χρόνια και στατιωτικοί και πολιτικοί φορείς χρησιμοποιούν τα διαστημικά συστήματα για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως επιτήρηση της γης, παρακολούθηση του περιβάλλοντος, έγκαιρη προειδοποίηση και αναγνώριση, πλοήγηση και επικοινωνίες. Τώρα όσον αφορά το Κοπέρνικος που είναι βασικός πάροχος στοιχείων για τη γη ε, σε όλο τον κόσμο που αναπτύχθηκε ε, δίνει μια επαρκή αυτονομία όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά χρειάζεται μια διαφανή διαχείριση, πρόθεση, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και περαιτέρω ανάπτυξη του όλου προγράμματος στις επόμενες γενιές. Η δυνατότητα να χειρίζεται κανείς πάρα πολύ μεγάλα ε, όγκο στοιχείων από ετερογενείς πηγές είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και εύχρηστη υπηρεσία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προστασία τη πρόσβαση στα δεδομένα για να προστατεύονται ευαίσθητε πληροφορίε. Η χρήση του Κοπένικο για λόγου ασφαλεία πιθανότατα ανάψει του ενδεχόμενου κινδύνου για το σύστημα και έτσι είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουμε σωστή προτεραιότητα όσον αφορά τα θέματα ασφαλεία για τι διαδικασίε και τα τμήματα του συστήματο. Όσον αφορά το Γαλιλαίο, που είναι το, δικό, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προηγήσεως για δορυφόρου, και το γεωστατικό σύστημα απλοήγησης το έγνος, που παρέχει υπηρεσίες και στις αερομεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές και χερσαίες επιχειρήσεις, ε, πρέπει να κινηθούμε ε, προς ε, μεγαλύτερη χρήση των διαστημικών στοιχείων από την αγορά και των υπηρεσιών και να χρησιμοποιούνται περισσότερο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να γίνεται αυτό μέχρι αναθεώρηση τη φυσάμενη νομοθεσία και να γίνεται ένα έλεγχο κατά πόσο η νομοθεσία ταιριάζει με τα διευθυντικά προγράμματα. Και αυτό πριν θεσπιστεί η νέα νομοθεσία. Έχουμε ένα παράδειγμα, το e-call και τον κανονισμό για τον ψηφιακό ταχογράφο. Οπότε χρησιμοποιούμε περισσότερο το GNSS ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, υποχρεωτική χρήση του συστήματος. Θέλουμε να έχουμε πλήρη κάλυψη από το έγκνο και θα πρέπει και η δυτή δυνατότητα του Γαλιλαίου να αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον. Θέλουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και δυνατότητα κρυπτογράφηση. Ταυτόχρονα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού δορυφορικού βιομηχανικού τομέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, είναι ισχυρή, να έχει ισχυρή βάση για διαστημική τεχνολογία και την κατάλληλη βιομηχανία ούτω ώστε να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, να αναπτύσσουμε, να εκτοξεύουμε, να λειτουργούμε και να εκμεταλλευόμαστε διαστημικά συστήματα να έχουμε τεχνολογική αυτονομία, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων και επίση να λαμβάνουμε υπόψη διάφορε σχετικέ πτυχέ. Χρειάζεται ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα Ευρώπη και γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένε δράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λύσουν τα προβλήματα ασφαλεία και άμυνα. Έτσι η Ευρώπη θα έχει πρόσβαση στο διάστημα ακόμα και στην περίπτωση κρίση. Καλωσορίζω το αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει διάφορε δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη για το διάστημα και την ενίσχυση τη χρήση των καινοτόμων συστημάτων ε, προκήρυξη διαγωνισμών για να τονώσουμε έτσι και την οτομία και να διερευνήσουμε νέε προσεγγίσει για να χρησιμοποιούμε ιδιωτικέ επενδύσει και συμπράξει με τη βιομηχανία. Άρα συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και θα πρέπει αυτό να γίνεται μέσω συμβάσεων ή μέσω ε, διαφόρων κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών, GTIs. Το GTI που πρότεινε ο κ. Μαρινέσκου Εδράζεται επί των πιλωτικών του προγραμμάτων και καινοτόμων δυσμικές τεχνολογίας ε, για να χρησιμοποιούμε καινοτόμα υλικά στο διάστημα, αλλαγή ε, τροχιά κλπ. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα να αυξήσει ο τομέα την ανταγωνιστικότητα και θα χρησιμοποιούνται οι, ε, για τι συμπράξει αυτέ δημόσιοι πόροι. Ένα μελλοντικό τέτοιο GTI μπορεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή για να καλύψει και μελλοντικέ ανάγκε. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια. Η στρατηγική υποδομή για το διάστημα είναι κάτι που απειλείται, διότι τα διαστημικά συστήματα απειλούνται πολλαπλώς. Από συγκρούσεις με απόβλητα κινδυνεύουν και άλλα διαστημικά αντικείμενα. Επίσης έχουμε και καιρικά φαινόμενα στο διάστημα, ε, μπλοκάρισμα διαφόρων εκπομπών, ε, επιθέσεις μέσα του κυβερνοχώρου και ίσως να υπάρχουν και επιθέσεις από αντιδορυφορικά συστήματα. Θα πρέπει τελικά να μην υπονομεύσουμε το, το χώρο του διαστήματος μέσω λαθασμένης συμπεριφοράς. Πρέπει να ανταποκριθούμε στι απειλές. Χρειαζόμαστε πολλά εργαλεία. Οι απειλές και απαντήσεις αυτές μοιάζουν για όλους όσους ανακατεύονται το διάστημα. Και από τον πολιτικό και τον εμπορικό και εξωτικό τομέα. Άρα χρειάζεται κοινή αντίληψη για τις απειλές. Μπορεί να είναι βάση για να βρούμε κοινέ απαντήσεις. Η ευρωπαϊκή διαστημική κοινότητα θα μπορούσε να αφοληθεί από κοινή στρατηγική και προβληματισμό. Έτσι μπορούμε να είμαστε πιο και όσον αφορά τι απειλέ κατά των συστημάτων μα. Να μην εξαρτώμεθα τόσο από εξωτερικού φορεί και μπορούμε να βοηθήσουμε ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο ασφαλέ ε, περιβάλλον για διαστημικέ δραστηριότητε. Η ανάπτυξη του συστήματο ανείχνευση και εποπτεία ε, του διαστήματο SST για να έχουμε ευαισθητοποίηση όσον αφορά το θέμα του διαστημικού χώρου, το SSA, αυτά τα δύο συστήματα βελτιώνουν την εποπτεία του διαστημικού χώρου. Χρειάζεται αποτελεσματική προστασία των δυστημικών μας μηχανισμών. Άρα, τα θέματα ασφαλείας θα πρέπει συμπεριλαμβάνονται όταν σχεδιάζουμε στρατηγικές, πολιτικές, την τεχνολογία και όταν παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις των δυστημικών προγραμμάτων, από σύλληψη μέχρι λειτουργία. Το 2016 είναι κρίσιμο έτος για την ασφάλεια του διαστήματος στην Ευρώπη. Οι αρχικές υπηρεσίες του Γαλιλαίου θα ξεκινήσουν. Το Κοπέρνικος μαζί με αποστολές θα συμβάλλει στην παροχή δεδομένων που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για ασφάλεια και άμυνα. Το consortium SST θα επεκταθεί. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική σε παγκόσμιο επίπεδο, η εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλεια ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για την άμυνα ούτω ώστε να εκμεταθεί και να ενισχύσει συνέργειες μεταξύ ασφαλείας και άμυνας, κυρίως στον τομέα του διαστήματος. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει νέα στρατηγική διαστημική για την Ευρώπη και η ΕΖΑ αναμένει να δημοσιεύσει μια νέα πολιτική για την ασφάλεια στο διάστημα. Πρέπει να υπάρχει κοινό στρατηγικό προβληματισμό για την ασφάλεια στο διάστημα. Έτσι μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε, να ανοίξουμε δρόμο για περαιτέρω επιχειρήσει στο μέλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια ανάγκη να συνεχίσει διάλογο με στρατηγικού διεθνεί εταίρου αφορά το διάστημα. Να χρησιμοποιήσουμε οικονομική διπλωματία και εμπορική πολιτική και έτσι θα ανοίξουν νέες αγορές για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και προβλήματα. Ήμουν συντομότερος από 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέροντα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Και τώρα περνούμε στις ερωταποκρίσεις. Κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τόρτορο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που επισημάνατε, το θέμα της ανταγωνιστικότητας, τόσο για τον κλάδο όσο και για τον πολίτη βέβαια. Για μένα αυτό σημαίνει ότι θα έχουν και οι πολίτες και τα θεσμικά όργανα πρόσβαση σε υπηρεσίες, στις ίδιες σε περισσότερες ακόμη, όπως και σε άλλους τομείς. με ένα υψηλό επίπεδο ποιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια είναι η δική σας γνώμη. για τον ανταγωνισμό με άλλες ζώνες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα κτλ. και τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε τους ε, δορυφόρους μας. Γιατί έχουμε δορυφόρους, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται κιόλα κατά τρόπο αποτελεσματικό. Και επίσης, έκανε λόγο και για την ε, διερεύνηση ο κύριος Τόρτορα. Εσείς που έχετε φτάσει εκεί ψηλά, τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουν αυτές οι δραστηριότητες στο διάστημα. Γιατί δεν νομίζω να προβλέπετε τίποτα για το μέλλον. Και θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο, χρήσιμο και ενδιαφέρον να αναπτυχθεί μια τέτοια δραστηριότητα ή όχι. Γιατί για μένα θα ήταν βέβαια χρήσιμο ή τουλάχιστον να αναπτυχθεί περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόχιτσεκ. Δύο ερωτήσεις. Η ανταγωνιστικότητα καταρχάς να είναι πολύ ε, σημαντική και απαραίτητη. Και θέλω να ρωτήσω τι άλλα στοιχεία χρειάζεται να έχουμε για να εκτοξεύουμε και να παρακολουθούμε τους δορυφόρους. Στοιχεία δηλαδή τα οποία χρειαζόμαστε όπως πυράβλους, εκτοξευτές, ε, σταθμούς εδάφους. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, ε, θέλετε να εκμεταλλευτείτε το εξοδιάστημα, δηλαδή πέραν των δορυφόρων, το χώρο πέραν των δορυφόρων, για να διερευνήσουμε άλλους πλανήτες ε, του ηλιακού μας συστήματος κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας παρακαλέσω τον κύριο Τόρτορα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής ε, Διαστημικής Πολιτικής πόσο έχετε συνεργασία στο πρόγραμμα Horizon 2020, σε ποιο βαθμό έχετε συνεργασία και επίσης γιατί το Horizon 2020 είναι γενικό μένα, μας εξασφαλίζει όμως βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Γιατί όταν παρακολούθησα τις ε, διαφάνειες και τις ε, σα Μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και θέλω να ρωτήσω το εξή. Ένα άλλο θέμα λοιπόν είναι ότι η πρόσβαση στο έδαφος, στο διάστημα εξαρτάται από το να μετατραπεί μια κυβέρνηση σε καταναλωτή. Εσείς λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε να, ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι θα γίνουν καταναλωτές αυτής της τεχνολογίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τι επίπεδο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Και κάτι ακόμη. Πρέπει να υποστηρίξουμε μια ιδέα τέτοια. Αυτή είναι ερώτηση προς ε, φόντερους τους ομιλητές μας γιατί είναι πολύ σημαντική. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικέ επενδύσεις για το διάστημα μέσω του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αυτό και για τους δύο μιλητές μας, και ιδιαίτερα για τον κύριο Κουνάριου, τον ε, προσκεκλημένο μας από την Ρουμανία. Ο Γιονκέρ έχει κάνει προτάσεις και για την άμυνα της Ευρώπης, ε, βελτίωση και του δυναμικού, του διαστημικού για λόγους ασφάλειας και προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το κρίνετε σε αυτό, τη δυνατότητα δηλαδή χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων. Και τρίτη ερώτηση, ποιες είναι οι βασικές απειλές που βλέπετε για την Ευρώπη από το διάστημα απειλές. Ή τεχνικής φύσεως, ή πολιτικής, ή οικονομικής βεβαίως. Γιατί λεφτά ποτέ δεν υπάρχουν αρκετά. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις των συναδέλφων και οι δικές μου. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Για τον κύριο Μαρινέσκου πρώτα. Δεν βλέπω γιατί πρέπει η Ευρώπη να οχριά σε σχέση με αυτό το οποίο προσφέρει αυτή τη στιγμή ως αποτέλεσμα. Στο χώρο του διαστήματος η Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι έχει χέρι ιδιαίτερου κύρους και αναγνώριση στη διεθνή σκηνή είτε λόγω των επιτευγμάτων της, στην ε, επιστήμη του διαστήματος, ε, στους, ε, στα παρατηρητήρια, τους εκτοξευστές με την Αριάν, κάθε τομέας δηλαδή. Σχετικό με το διάστημα. Και μάλιστα θα το έλεγα αλλιώ ότι το διάστημα είναι από τους λίγους τομεί υπεροχή της Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με του άλλου ανταγωνιστέ. Και μάλιστα έχει καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα η Ευρώπη δαπανώντας κλάσμα μόνο αυτών που έχουν δαπανήσει οι ανταγωνιστές της. Δεν βλέπω κανένα λόγο, λοιπόν, να αμφισβητεί κανείς την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα αυτών. Σε σχέση με την διερεύνηση, αν θα πρέπει η Ευρώπη να δραματίσει ρόλο στη διερεύνηση. Ναι, συχνά ακούμε να λένε «Α, δεν είναι στιγμή κατάλληλη, οικονομική κρίση» κτλ. κτλ. Θα σας απαντήσω ως εξής, ότι αν περιμένουμε να έρθει η στιγμή που θα μας περισσεύουν τα λεφτά και δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν θα παίξει ρόλο στην διερεύνηση του διαστήματος η Ευρώπη, προφανώς δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Τώρα ίσως θα πρέπει να δούμε το ερώτημα αντίστροφα. Έχει περιθώριο και οικονομικό η Ευρώπη να παραμείνει απούσα, απολύτως απούσα από το μέλλον και τις διεθνείς συνεργασίες που αναμφίβολα θα αναπτυχθούν. Αναμφίβολα γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνημα για την ε, διερεύνηση του ηλιακού συστήματός μας αλλά και πέραν αυτού. προσωπική μου λοιπόν ε, θέση είναι ότι η Ευρώπη που έχει τη φιλοδοξία να είναι μια κοινωνία και οικονομία στηριζόμενη στη γνώση πρέπει, οφείλει να διαδραματίσει ρόλο. Άρα πρέπει να ορίσουμε, πιστεύω, φιλοδοξίες που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχουν. Τώρα, το SST και γενικά παρακολούθηση των εξελίξεων στην ε, εγκύτερη, στην ε, γη τροχιά. με βάση και τις ε, τοποθετήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έγγραφο για το πρόγραμμα SST, βλέπουμε ότι είναι αξιέπαινες οι προσπάθειες. το SST, Space Surveillance and Tracking, είναι η προσπάθεια να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν τεχνικά από το έδαφος με βάση την υπόθεση πώς θα αξιοποιούνται εκτεταμένα τα συστήματα παρακολούθησης από εδάφους για να βλέπουμε τι συμβαίνει στο έστωμα, αλλά και αυτό έχει τα όρια του. Και στο τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να ανοιχνεύσουμε και στο πώς μπορούμε να ορίσουμε πρόσβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη γνώση σε σχέση με τα μικρότερα αντικείμενα του διαστήματος αυτά δηλαδή, τα οποία δεν ανοιχνεύονται από εδάφους. Άρα υπάρχει μετά το SST ένα επόμενο βήμα που είναι το SSA τα εσωτερικά συστήματα ανείχνευσης από το διάστημα δηλαδή που ανοιχνεύουν τα απόβλητα, τα διαστημικά απόβλητα, γιατί έχουμε διαρκή παραγωγή αποβλήτων, πολύ ταχύτερη από ότι ε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε σχέση με αυτά που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα. Και ως εκ τούτου πρέπει να μας απασχολεί το θέμα. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Αυτή τη στιγμή στηριζόμαστε στο δυναμικό των ΗΠΑ και χωρί να υπάρχει κανένα λόγο να το αποκλείσουμε αυτό, να στηριζόμαστε δηλαδή στο δυναμικό των ΗΠΑ για την παρατήρηση του διαστήματο, ερωτώ πόσο θέλουμε να είμαστε τυφλοί. Ερώτηση μόνο, γιατί απάντηση δεν έχω. Αλλά πάντω είναι μια ερώτηση στην οποία πρέπει να δοθεί απάντηση κάποια στιγμή. Για τον κύριο Μπούζεκ και τον ορίζω το 2020. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε ε, συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό, ορίζον 2020 και ανταγωνιστικότητα και θα ήθελα εν προκειμένου να χαιρετήσω τις ε, προσπάθειες στις οποίες αποδιέται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει απαντήσεις, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κλάδου Αλλά εν νομίζω ότι έχουμε ζήτημα ε, διακυβέρνησης του προγράμματος. Και πρέπει να προσδιοριστούν και οι στόχοι, να γίνουν οι επιλογές και, και να οριστούν οι προτεραιότητες για τις δραστηριότητες κτλ. Καταναλωτής ή πελάτης. Άλλη ερώτηση. Βεβαίως πολύ ενδιαφέρουσα και θα δώσω δύο απαντήσεις. Πρώτον, ότι αν το SpaceX ήταν πρόγραμμα της NASA, τον προπολογισμό της NASA θα τον είχε ψηφίσει μόνο η Καλιφόρνια. Για το SpaceX στηρίζεται στην περιορισμένη καινοτομία και τη ριζική βελτιστοποίηση της επανοργάνωσης του κλάδου, δηλαδή συγκέντρωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε ένα μόνο τόπο, την Καλιφόρνια. Καμία αναδιανομή δηλαδή δραστηριοτήτων ή κατανομή δραστηριοτήτων μεταξύ των πολιτιών, και ασφαλώς στην υποθετική αυτή περίπτωση το πρόβλημα αυτό δεν θα μπορούσε να έχει υλοποίηση και χρηματοδότηση δημόσια. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Γι' αυτό και από την έννοια του πελάτη περάν στην έννοια του καταναλωτή και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το SpaceX. Και τις οποίες είναι διατεθειμένος να αγοράσει ο καταναλωτής. Εμείς στην Ευρώπη απέχουμε πολύ από αυτή την θεώρηση και την προσέγγιση, χωρίς να λέω ότι πρέπει να αντιγράψουμε το μοντέλο SpaceX, το Ariane 6 παραδείγματι. Είναι καλός τρόπος, είναι μια ουσιαστική εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση, παραμένει ωστόσο σε εμβιβαστική. Θα δούμε βέβαια και θα αποφασίσει η αγορά εάν είναι ικανοποιητικός αυτός ο συμβασμός ή όχι. Είναι νωρίς νομίζω ακόμα. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις θετικές επενδύσεις. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, το είπα και νωρίτερα. Ας εκθέσω μερικές. Πρώτον, πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο επιδόσεων. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα και οι δεσμεύσει μακροχρόνια. Να δώσω το παράδειγμα του Γαλιλαίου, αν μου επιτρέπετε. Εάν αναλογιστείτε ότι κάθε φορά που το Γαλιλαίο αντιμετωπίζει δυσκολίε και δυσκολίε υπάρχουν, ασφαλώς και υπάρχουν ε, πάντα, απρόβλεπτα εμπόδια, δυσκολίες τεχνολογικές, ε, αποτυχίες κατά την εκτόξευση, τεχνικές δυσκολίες. Κάθε φορά που τα βλέπουμε αυτά, κάποιος αμφισβητεί το πόσο απαραίτητη είναι η επένδυση. Να σας δώσω το παράδειγμα του GPS και το GPS και τεράστιες δυσκολίες, κατά πάσα πιθανότητα πολύ περισσότερες από ό,τι έχει ε, αντιμετωπίσει το Γαλιλαίος. Ακούσατε ποτέ κανέναν να αμφισβητεί την ε, χρησιμότητα του GPS από πλευρά των ΗΠΑ. Ούθεις. Και αυτό είναι το όνειρό μου κάποια μέρα οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν μια ξεκάθαρη δήλωση για το Γαλιλαίο, να πούνε ναι, μπορεί να περνάει από κάποιε δυσκολίε μεν, αλλά θα υλοποιηθεί όσο και να χρειαστεί, όσο και να κοστίσει αυτό. Αυτό θα ήταν μια τεράστια ε, σημασία κίνηση και θα καθησίκαζε και τους επενδυτές. Και εδώ και το θέμα των ε, της ασφάλειας και των υποδομών. Έχει τεράστια ε, σημασία για να γεννώνται πολλά ερωτήματα και από τα απόβλητα τα διαστημικά όπως είπαμε αλλά και για άλλες νέες απειλές που προκύπτουν και οπωσδήποτε πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό σημαίνει μια σειρά από εξελίξεις και ρυθμιστικές παρέμβασεις νομοθετικής, διάλογου διεθνούς, δεν μπορεί δηλαδή εσωτερικά μόνο να διευθυνθεί και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον παραλυσμό ως προς το κυβερνοχώρο και το διάστημα. Τα δύο αυτά άειλα διαστήματα που έχουν τόσο μεγάλη σημασία τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με αγαθό κοινό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αγαθά τα οποία χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες του κόσμου. Και δεύτερον, δύο διαστήματα, κυβερνοχώρος και διάστημα, όπου δεν υπάρχει σύστημα διακυβέρνησης διεθνές. Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, Δεν πρόκειται για τον κυβερνοχώρο, δεν πρόκειται για το διάστημα. Δεν υπάρχουν ε, εθνικές διατάξεις ή δεν υπάρχουν γενικώ ρυθμίσεις. Και κανείς δεν θα μιλήσει αν η ελάχιστοι κανόνες της ε, αυροφροσύνης, της ορθής συμπεριφοράς κτλ. παραβιάζονται. Ξεκάθαρο αυτό. Και επίσης τρίτο εξυγχρονισμός. Και στις δύο περιπτώσεις. Αυτά είναι τα τρία παράλληλα χαρακτηριστικά των δύο χώρων, του κυβερνοχώρου και του διαστήματος, που ήθελα να σας παρουσιάσω για να αντιληφθείτε τη σημασία. Για το κυβερνοχώρο ίσως τον βλέπουμε, τον κατανοούμε περισσότερο καθώς είναι πιο κοντά στην καθημερινή μας ζωή. Το ίδιο ισχύει όμως και για το διάστημα. Και η κατάσταση είναι μάλλον ανησυχητική αυτή τη στιγμή. Αυτά ως προς τις βασικές μου ιδέες και απαντήσεις. Το σεληνιακό χωριό. Α, νόμιζα ότι το κάλυψα, γιατί είχε να κάνει με τη διερεύνηση, μελλοντικές εξελίξεις και δυνατότητες ανάπτυξης. Πέραν του ΑΕΣΕΣ, η σελήνη θα είναι το επόμενο λογικό βήμα, πιστεύω, μετά το ΑΕΣΑΣ. Τώρα θα είναι σιλινιακό χωριό, θα είναι κάποια υποδομή περί, το, περί Ε, είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Πρόεδρε, η σειρά μου. Διαρεύνηση πρώτα απ' όλα. Η διερεύνηση σημαίνει γνώση και πρόοδο, πιστεύω. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει πίσω στην αναζήτηση γνώσεως και πρόοδου σε σχέση με το διάστημα. Το να γνωρίζουμε περισσότερα για τα ηλιακά συστήματα, για τους αστέρες, τους γαλαξίες, σημαίνει να γνωρίζουμε και καλύτερα πώς έχει διαμορφωθεί η γη, πώς έχει προκύψει η ζωή και άρα μπορούμε και να προβλέψουμε καλύτερα το τι μπορεί να συμβεί για μας, για τον πλανήτη μας στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή θα έχετε δει ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον, για ε, Άρη. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ίσως εκατομμύρια χρόνια, μπορεί να υπήρξε νερό από ό,τι φαίνεται στον Άρη. Αυτό αποδεικνύεται από τη διάβρωση του εδάφους τι συνέβη στον πλανήτη αυτό. Αυτό πρέπει να μάθουμε για να καταλάβουμε τι συνέβη στον Άρη και να αποφύγουμε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στο δικό μας πλανήτη. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε τη διερεύνηση του διαστήματος. Ταυτόχρονα είναι πολλοί οι κίνδυνοι που προέρχονται από το εξοδιάστημα διαστημικές καταγίδες, σε παραδείγματι, που μπορεί να επηρεάζουν την ηλεκτρονική τεχνολογία των δορυφόρων, τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, πολλές φορές ακόμη και, τις, και τους αεροδιαδρόμους που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα, Κοστίζει χρόνο, κοστίζει χρήμα. Πρέπει να γνωρίζουμε χάρη στη ερεύνηση λοιπόν του διαστήματο και του εξωδιαστήματο τι σημαίνουν τα φαινόμενα αυτά, τα καιρικά φαινόμενα του διαστήματο, να τα μελετήσουμε και να αναπτύξουμε τα τεχνικά εκείνα μέσα που θα μα επιτρέπουν να αποφύγουμε τι συνέπειές του στις δυσμενείς στο μέλλον. Αστεροειδείς που επίσης αποτελούν κίνδυνο για τη Γη. Αν αναλογιστούμε το 1908 ο αστεροειδής των Γκούστα ε, εκρίζωσε 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με συνέπειες ιονισμού που φτάσανε μέχρι τις βόρειες χώρες Σκανδιναβίας και τη Βρετανία με 4-5 μέτρα διάμετρο μόνο. Το, το 1914 στο Τσαργκάνιστ, στα Βαλκάνια κοντά, όχι τόσο μακριά, έπεσε αστεροειδής με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάνια σε ολόκληρη την πόλη, να ξυριστούν ορισμένα ψηλά κτίρια, να χάσουν τη ζωή τους περίπου τους 300 πολίτες. Ε, τώρα προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το πώς είναι αυτά τα φαινόμενα των αστεροειδών. Μια πτυχή που σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών τώρα έχει, μελετάται πολύ με δύο χωριστούς φορείς, Διεθνές Δίκτυο Αστεροειδών και Συμβουλευτική Ομάδα για το Σχεδιασμό του Διαστήματος. Σημαντικές διαστημικές υπηρεσίες δε, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, συμμετέχουν στα δίκτυα αυτά, πράγμα που σημαίνει διερεύνηση, μελέτη και εφαρμογές και για τη γη. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο. Αλλά θα πω ότι διαρεύνηση σημαίνει πάνω απ' όλα συνεργασία. Πρώτα απ' όλα συνεργασία. Γιατί ε, έχει να κάνει με τα προβλήματα που αφορούν την υφήλιο, τον πλανήτη Γη. Άρα, η συνεργασία μεταξύ των μεγάλων υπηρεσιών του διαστήματος με κονδύλια πολύ περισσότερα από, τα, όσα μπορεί μία μόνο αποστολή να καλύψει, δηλαδή χωριστά οι ΗΠΑ, η Κίνα ή όποιος άλλος. Γιατί σημαίνει ταυτόχρονα συνεργασία ηλικείται και ε, Και αυτό μπορεί να σημάνει και την ειρήνη για ορισμένα ζητήματα που απασχολούν τις χώρες μας. Αν σκεφτούμε την γη ως ένα σύνολο. Το σεληνιακό χωριό. Βεβαίως μπορεί αυτό να δώσει απαντήσεις για τη διερεύνηση. Μπορεί επίσης να δώσει απαντήσεις για μελλοντικά ωφέλη που θα μπορούσε η Ευρώπη να υπολογίζει πώς θα εξασφαλίσει. Φερρυπίν. Υπάρχουν πολλοί φυσικοί πόροι στη σελήνη. Μπορούν να αξιοποιηθούν. Και σε κάποιο πλαίσιο ίσως θα ήταν και πιο ε, ευχερές και φθηνό να γίνεται η εξόριξή τους στην σελήνη και όχι στη γη. Το υδρογόνο 3 επί παραδείγματι που ορισμένοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αξιοποιήσουν ως πηγή ενέργειας. Μπορούμε να το αντλήσουμε από τη σελήνη και μετά τη σελήνη και από, από άλλους πλανήτες. Το ελληνικό χωριό βέβαια αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα εγχείρημα, δεν είναι ένα υπαρκτό έργο. Αλλά πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να αντιληφθούν την αναγκαιότητα, να πάμε πέρα από αυτό, να διερευνήσουμε, να φτάσουμε στο επίπεδο της γνώσης που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Να κοιτάξουμε λοιπόν το πρώτο ουράνιο σώμα, το πιο κοντινό στη Γη. 380.000 χιλιόμετρα μόνο απέχει από, την, από τον πλανήτη μας. Αυτό είναι η δική μου θεώρηση, η δική μου σκοπιά σε σχέση με το σεληνιακό χωριό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η, η κάλυψη των αναγκών σε άμυνα από το Ταμείο του κ η Ευρώπη, όπως κάθε άλλο, η οντότητα επιγής που ασχολείται με, τον, με το διάστημα, αντιμετωπίζει απειλές από διάφορους παράγοντες, είτε εξωτερικούς, όπως είπα, διαστημικές καταιγίδε, αστεροειδείς και ούτω καθεξής, αλλά και ανθρώπινους παράγοντες. Επίθεση από πιθανούς εχθρούς, όχι η κράτη αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η τρομοκρατία, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονό ότι αργά ή γρήγορα θα έχουν τη δυνατότητα τη πρόσβαση στο διάστημα οι τρομοκράτε, γιατί κάποιοι από αυτού έχουν αρκετό χρήμα και αρκετή γνώση επιστημονική για να προαγάγουν τέτοια εγχειρήματα και να φέρουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ευρωπαϊκά συστήματα, αλλά και συστήματα άλλων κρατών. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις, τις νέες απειλές, όπως και τις κυβερνοαπειλές επίσης. Όσο πιο πολλά χρήματα λοιπόν διαθέσουμε στα αμυντικά συστήματα με την προαγωγή της ασφάλειας και της άμυνας, τόσο το ταχύτερο θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Και δεν πρέπει να λεσμονούμε ένα πράγμα. Ότι διαχρονικά η ανάπτυξη του διαστήματος σε χώρες όπως η Ρωσία, πρώην Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε, μεταξύ των δύο αυτοκρατών, ξεκίνησε πρώτα από το στρατιωτικό σκέλος με στόχο τη διασφάλιση όχι μόνο τη κλίνηση μιας δομής και την ασφάλεια ενό συστήματος, αλλά και την ασφάλεια ενό συστήματος. Η Ευρώπη έμεινε πίσω σε όλες αυτές τις πτυχέ η Ευρώπη ξεκίνησε τα προγράμματα έχοντας υπόψη τον πολίτη, τις εφαρμογές για την καθημερινή ζωή και μετά άρχισε να την απασχολεί το ζήτημα της ασφάλειας των ε, συστημάτων της. Τώρα αρχίζουμε να ε, προσεγγίζουμε αυτή τη ε, διάσταση και να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτήν. Ευπρόσδεκτε όλε οι πρωτοβουλίε για μένα. Α προσπαθήσουμε όλε αυτέ τι πτυχέ να τι εντάξουμε σε μια κοινή στρατηγική, σε ένα κοινό εγχείρημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε για να μάθουμε τόσα για το διαστημικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέρφους, τους βοηθούς, τους συμβούλους που ήταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε στην Ήτρε στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Σύντομα δηλαδή σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω όλη η μελλοντική εξερεύνηση θα είναι επικοδομητική για την Ευρώπη, επιτυχής για την Ευρώπη. Και ευχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ.